Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Είμαστε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με τον Μάριο Μορκόνη, που είναι ο Ιταλς υπουργό Εσωτερικών, και τον Ζων Κριστόφο Φιλόρη, που είναι επικεφαλής τμήματάρχης δηλαδή του Τμήματος για το Μαγκρέπ στην Γενική Διεύθυνση ΝΙΕΡ και τον Βίνσεντ Πικέ που είναι και αυτός του για το Μακρέπ στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον Μάρτ Χίτεμαν που είναι από την Εστονική Προεδρία. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι. Οι συντονιστές αποφάσισαν το Σεπτέμβριο να καλέσουν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να παρουσιάσουν λεπτομέρειες για τις πρόσφατες εξελίξεις στο μεταναστευτικό ε, όσον αφορά τη Λιβύη. Και χαίρομαι λοιπόν που έχω εδώ πέρα τόσο εξέχοντες ε, προσκεκλημένους. Μιλάμε για τα hot spots ε, συχνά και για άλλα. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Μάριο Μορκόνη, Υπουργείο Υπουργείου Επαμεσωτερικών της Ιταλίας και μετά στους ε, επόμενους. Να είσαστε σύντομη παρακαλώ. Νομίζω ότι στη συζήτηση θα έχετε την ευκαιρία να πείτε περισσότερα. Οπότε και πάλι πολύ χαίρομαι που μπορώ να δώσω το λόγο στον ομάρχη κύριο Μάριο Μορκόνε από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι έχετε ξανάρθει εδώ και πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε και ευχαρίστως να σας ξαναέχουμε και σε άλλες ευκαιρίες μαζί μας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και για την ευκαιρία που μου δίνετε να εξηγήσετε ποια είναι η Ιταλική προσέγγιση στο θέμα αυτό που για μας είναι καθοριστική σημασία. Πρόκειται για τη σχέση με την Αφρική, κυρίως με τη Λιβύη. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Ιταλία. Ε, με την υποστήριξη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το θέμα έχει αναχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συζητήθηκε στη συνάντηση κορυφής ε, της Βαλέτα τη συνάντηση και με την Αφρική υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο προβλέπεται για τη χρηματοδότηση αυτής της σχέσης. Κατά τα άλλα και στην, ε, ε, στο, Υπουργείο, στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη στο Ταλίν τον Ιούλιο, πέρα από τις ε, διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν για διάφορα θέματα, όμως προέκυψε το ότι πρέπει να αναλυφθούν δράσεις οι οποίες συζητήθηκαν και πρόσφατα στο Παρίσι ε, με τον κύριο Βραμόπουλο και με τη Γερμανία. Η Ιταλία λοιπόν ε, θεωρώ ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο βέβαια και γεωγραφικής ε, σημασίας ε, όσον αφορά την κρίση της Μεσογείου. Στη Ρώμη εμείς ανακοινώσαμε ότι θα υπάρξει ένα φόρουμ πολιτικό, ομάδα επαφής κατά κύριο λόγο, πρόκειται για ομάδα επαφής με τις χώρες Αφρικής για το θέμα των μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο, κυρίως από τη Λιβύη και την Τινησία. Μετά από αυτήν την πρωτοβουλία, πέρα από το ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων, διαπιστώθηκε ότι και στη δεύτερη διάσκεψη στην Τινησία πριν από λίγους μήνες, οι υπουργοί ε, αποφάσισαν να συναντηθούν στην Πέρνη στις 13 Νοεμβρίου. Λιβύη, Μαλή, Νίγηρας, με αυτές τις χώρες έχουμε ιδιαίτερε επαφές. Και στις 28 ε, Αυγούστου ήταν η τελευταία συνάντηση, ε, θα ακολουθήσει στις 6 Δεκεμβρίου μια τεχνική τεχνική επαφή, τεχνική συνάντηση για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε πρακτικά για να αντιμετωπιστεί η νόμιμη μετανάστευση και γενικότερα μεταναστευτικέ ροές. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες. Η δική μας η στρατηγική, την οποία στηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να υπάρχουν τρεις άξονες. Πρώτος άξονας αφορά τους ε, διακινητές, δεύτερος ε, αφορά την ε, διαβίωση γενικότερα και το τρίτο αφορά την διάσωση στη θάλασσα, αλλά και το πώς μπορούν να βελτιωθούν ε, οι συνθήκες διαβίωσης ε, των μεταναστών που έρχονται από τη Λιβύη και από άλλες αφρικανικές χώρες. Η υποστήριξη προς τις ε, τοπικές κοινότητες και αυτό είναι κάτι που λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη. Όσον αφορά λοιπόν τους ερχόμενους από τη Λιβύη, ε, για να ε, διαχειριζόμαστε καλύτερα τα θαλάσσια σύνορα, αλλά έχοντας κατά νου και τα ε, πυρωτικά σύνορα, λαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εναντί των διακινητών να περιστούν και οι θάνατοι στη θάλασσα. Έχουμε λοιπόν μία μείωση των θανάτων αυτών κατά 32,5%. Εξάλλου πέρα από αυτά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε καθορίσει ένα πολιετές ε, πρόγραμμα που βασίζεται σε δύο σημαντικά σε δύο σημαντικές φάσεις. Η πρώτη είναι από το 17 μέχρι το 20. Εκεί προβλέπονται τέσσερις σημαντικές δράσεις. Η υλοποίηση λειτουργικών και επιχειρησιακών, επιχειρησιακών μάλλον κέντρων θα είναι ένα είδος ε, κέντρων συντονισμού. Εκεί θα γίνεται ο συντονισμός και για την θαλάσσια διάσωση. Ε, δεύτερη φάση θα αφορά στην γενικότερη διαχείριση της ασφάλειας ε, στις ακτές. Η τρίτη δράση είναι παροχή βοήθειας στην ακτοφυλακή της Λιβύης έτσι ώστε ε, να καθορίζεται και για αυτούς το πεδίο στο οποίο θα μπορούν να διασώζουν ζωές. Το τέταρτο αφορά να υπάρχει καλύτερη ε, διαχείριση των υπηρετικών συνόρων. Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα το διαχειρίζεται μια τεχνική επιτροπή και θα οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση των ε, υπηρετικών συνών. Αυτά για την πρώτη βάση. Η άλλη από το 21 μέχρι το 26. Εκεί θα είναι δράσεις που θα αφορούν και πάλι ε, στον συντονισμό των διαφόρων δυνάμεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. 280 περίπου εκατομμύρια θα είναι το κόστος όλης αυτής της δράσης. Τα κονδύλια θα έρθουν και από την Ιταλία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα στην, ε, στη, ε, στη συνεργασία με τη Λιβύη για θέματα μετανάστευσης, ε, έχουμε έξι συγκεκριμένα σκάφη τα οποία διαθέτουμε στην ακτοφυλακή της Λιβύης και μέχρι το τέλος του έτους θέλουμε στη Λιβύη να δώσουμε άλλα τρία σκάφη. Παράλληλα ε, οργανώνουμε στα δικά μας τα ειδικά κέντρα ε, σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού έτσι ώστε το προσωπικό να μπορεί να χειρίζεται τη σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να συντονίζεται και με τους άλλους ε, ειδικού ε, που ασχολούνται με τη ε, θαλάσσια διάσωση. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Υπάρχουν και άλλα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο προσπαθούμε να προγραμματίσουμε και την υποστήριξη που προσφέρεται στις τοπικές κοινωνίες τρίτων υπηκόων υπηκών από τρίτες χώρες. Ήδη προβλέπετε ότι θα ε, προσφέρουμε βοήθεια με τη μορφή τροφίμων αλλά και φαρμάκων. Οι συναντήσεις τις οποίες είχαμε με τους ε, δημάρχους ε, των λιβικών κοινοτήτων μας οδήγησαν σε ένα διάλογο από τον οποίο προέκυψε, προέκυψαν μία σειρά ε, δράσεων και μέτρων που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά ε, και κρίνουμε και επίση απαραίτητα. Είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν το θέμα των ποσοστώσεων. Ε, η Πρόκειται συγκεκριμένα για προγράμματα τα οποία αφορούν στην υποδομή, στην ασφάλεια, αλλά Πρόκειται επίσης και για προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο να προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στην οικονομία η οποία στηρίζεται στην παράνομη διακίνηση. Ε, πρέπει να βελτιωθεί η διαβίωση στις τοπικές κοινότητες και όχι μόνο αυτό αλλά να βελτιωθούν και οι υγειονομικές δομές, η συντήρησή τους, η υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων μπορεί και πρέπει να αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στην σταθεροποίηση της Λιβύης. Να ενισχυθούν οι θεσμοί και με τον τρόπο αυτό θα αναχαιτιστούν και οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Νομίζω όμως ότι αυτό που επίσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Επιτροπή είναι ο ρόλος των οποίο έχουμε αναλάβει και σε σχέση με τις ΜΚΟ. Όπως ε, ε, αναφέρθηκε ήδη, θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει, να αντιμετωπιστούν οι λάθροδιακινητές. Κυρίως ε, σε σχέση με τη Λιβύη, γιατί εδώ και χρόνια ε, υπάρχει αυτή η παράνομη διακίνηση. Εμείς λοιπόν ε, προσπαθούμε να ε, συνεργαστούμε με τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών που είναι καθοριστική σημασία για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε τους στόχους μας που είναι να γίνονται σεβαστές οι προδιαγραφές και κυρίως στα κέντρα υποδοχής. Υπάρχουν θετικά στοιχεία, ε, αυτά διαπιστώσαμε στην Επιτροπή Ιταλίας ε, Λιβύης, ε, καταλήξαμε στο ότι συμμεριζόμαστε τους ίδιους στόχους, αυτό το επιβεβαίωσαν και οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Έτρων που παρίσταντο και αυτοί στην συνάντηση αυτή. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επισκεφθεί πάρα πολλά κέντρα υποδοχής και παραμονής στην Λιβύη. Ε, πρέπει να υπάρξει διεθνής προστασία γιατί η κατάσταση είναι ευαίσθητη και να υπάρξει και μεταγκατάσταση σε άλλες χώρες. Να έχουμε ένα ανθρωπιστικό διάδρομο, έναν διάβλο που θα επιτρέψει να ε, βοηθηθούν, να υποστηριχτούν 9.000 επιστροφές προς τις χώρες προέλευσης. Εμάς λοιπόν μας ενδιαφέρει η συντονισμένη παροχή βοήθειας μαζί με τους δημάρχους των ελληνικών κοινοτήτων. Η διεθνής κοινότητα στηρίζει και αυτή τις προσπάθειες. Πριν από τρεις μήνες συναντήθηκαν οι αρμόδιοι Υπουργοί Εστερικών και υπουργοί, Υπουργός από την Λιβύη και υπέγραψαν μια δήλωση δεσμευστική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος είναι ε, το να υπάρξει βοήθεια οικονομική από την Ευρώπη και από τη δική μου τη χώρα. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η πρεσβεία μας στην Τρίπολη γιατί διαμεσολαβεί και με τις, στις επαφές με την ε, Λιβύη. Ο ρόλος των ΗΠΑ είναι και αυτός καθοριστικής σημασίας για τις σχέσεις ε, με την Βόρεια Αφρική. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορά πολλές αφρικανικές χώρες και τη Λιβύη. στη Λιβύη πιο συγκεκριμένα σε πρώτη φάση που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου η ύπατη αρμοστή αποφάσισε να διεξάγει σεμινάρια για περίπου 150 υπαλλήλου έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί παράνομη η παράτυπη μετανάστευση ε, να γίνουν ε, σεμινάρια για, για τις προϋποθέσεις χωρίς ασύλου μαζί με την ε, κυβέρνηση της Τρίπολης θελήσαμε να καθορίσουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές για αυτά τα σεμινάρια, κυρίως όσον αφορά την, τα κέντρα υποδοχής. Ε, με αυτές τις πρωτοβουλίες ε, 283 ε, κρατούμενοι στα κέντρα απελευθερώθηκαν, αφέτηκαν ελεύθεροι. Επίσης υπήρξαν και πάρα πολλές άλλες ε, παρεμβάσεις σε πρώτο και σε δεύτερο επίπεδο, επεμβάσεις γιατρών ε, στα κέντρα υποδοχής, γιατί θελήσαμε να κρίνουμε το πώς ακριβώς διαβιούν περίπου 1980 άτομα σε αυτά τα κέντρα. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος, είπα τη ε, αρμοστία των προσφύγων καθόρισε και άλλες διόδους για να μπορούν να επωφεληθούν 400 περίπου πρόσφυγες που είναι πιο ευαίσθητοι και βρίσκονται στη Λιβύη. Αυτό το πρόγραμμα ε, θα προβλέπει και την ε, ε, προαιρετική τους και με δική τους βούληση επιστροφή στις χώρες προέλευσής τους. Οι ευαίσθητες ομάδες, οι γυναίκες και τα παιδιά μεταφέρθηκαν τον προηγούμενο μήνα στο Νίγηρα και από εκεί θα μεταφερθούν σε άλλες χώρες ε, οι οποίες θα είναι πρόθυμες ε, να τους ε, δεχτούν μέσα από την μετεγκατάσταση. Περίπου χίλιες θέσεις προβλέπονται πάντα αυτό το οργανώνει η ύπατη αρμοστία των προσφύγων, χίλια άτομα να μπορούν να φιλοξενηθούν άτομα τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση και τα οποία χρήζουν διεθνού προστασίες. Η δική μου χώρα προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί στην περιοχή για να ε, μπορέσει η αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών να έχει την απαραίτητη βοήθεια έτσι ώστε και αυτή να προσφέρει καλύτερα την ε, προστασία που επιθυμεί να προσφέρει. Θέλω να πω, εύχομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Είπα αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών ε, θα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο εκπρόσωπος ε, σε αυτή τη συνάντηση θα είναι ο κύριος Σαλαμέ. Ε, επίσης θέλω να επισημάνω ότι ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών στη Λιβύη για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες. Στους πρώτους εννέους μήνες οργανώσαμε πάντα με την υπατιαρμοστία την εκπαίδευση υπαλλήλων της ακτοφυλακής ε, γιατί στόχος μας είναι η αναδιάρθρωση των σημείων όπου γίνεται η απόβαση των μεταναστών να βελτιώσουμε τα κέντρα υποδοχής. Ε, Επίση, ε, διανύμουμε και σε πάρα πολλούς αποδέκτες αντικείμενα και τρόφιμα και φάρμακα τα οποία χρειάζονται. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ολοκληρώσω και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας ε, εφόσον το κρίνετε απαραίτητο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μορκόνε. Πολύ θέλω το λόγο για αυτό το σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας, οπότε σας παρακαλώ τους επόμενους ομιλητές να είσαστε συνοπτικοί γιατί θα ακούσουμε πολλές ερωτήσεις οπότε πολλά θα μπορέσετε να πείτε και στις απαντήσεις που θα δώσετε. Οπότε περιοριστείτε στα εμβλητικά σημεία της παρουσίασής σας. Οπότε περνάμε τώρα στον κύριο Ζαν Κριστόφ Φιλόρη που είναι προστάμενος της μονάδας Μαγκρέμπ στην Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση. 5 με 10 λεπτά παρακαλώ. Πρόεδρε, καλημέρα. Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, καλή σας μέρα. Μια υπόσχεση πρώτα. Δεν θα σας πλημμυρίσω με νούμερα. Όμως, θα σας δώσω μια συνολική εικόνα των προσπαθειών που κάνουμε εμείς μέσω του καταπιστευματικού ταμείου για την Αφρική και πιο συγκεκριμένα για τη Βόρεια Αφρική που καλύπτει και το πρόγραμμά μας για την Λιβύη. Στην Λιβύη έχουμε επί του παρόντος πρόγραμμα αξίας 162 εκατομμυρίων ευρώ. Τα τρία τέταρτα του ποσού αυτού πάνε στην προστασία των μεταναστών και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κοινοτήτων υποδοχής αυτών των μεταναστών. Το 1 τέταρτο του ποσού αυτού θα πάει σε δράση κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων των ακτοφυλάκων στη Λιβύη, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πιο ανθρώπινη διαχείριση, πιο επαγγελματική της μετανάστευσης σε αυτή τη χώρα, στη Λιβύη. Όσον αφορά την προστασία, υπάρχουν διάφορες δράσεις μέσω των εταίρων μας επιτόπου που είναι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Πατιαρμοστία αρμοστία για τους μετανάστες, αλλά και η UNICEF, αλλά και το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Όπως επίσης και η Γερμανική Αναπτυξιακή Οργάνωση και η Κατά πρώτον, λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει η βοήθεια στους μετανάστες εκεί όπου φτάνουν με ιατρική περίθαλψη και με ψυχική και κοινωνική υποστήριξη. Υπάρχει επίσης ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες, στους καταβλισμούς, στα κέντρα όπου συγκεντρώνονται. Βοηθούμε τους μετανάστες Δυστυχώς κάτω από συνθήκε που είναι πραγματικά απέσιες και γι' αυτό και επικεντρωνόμαστε στη βελτίωσή τους. Η δράση της προστασίας καλύπτει επίσης και τον επαναπατρισμό για ανθρωπιστικούς λόγους, των πιο ευάλωτων περιπτώσεων. Από την αρχή της χρονιάς, χάρη στη δικιά μας στήριξη, μπόρεσε ο ΑΕΜ να στηρίξει 10.000 μετανάστες προκειμένου να επιστρέψουν και ο στόχος των 15.000 θα επιτευχθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Είναι σαφές ότι μία από τις κύριες προτεραιότητές μας για του χρόνου θα είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή τη δράση μέσω του καταπιστευματικού ταμείου για την Αφρική. Η δράση τώρα στις κοινότητες υποδοχής στηρίζει τις τοπικές κοινότητες στη Λιβύη προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη μαζική αυτή ροή μεταναστών που βαραίνει κακά τα ψέματα πολύ πάνω σε αυτές τις τοπικές κοινότητες. Η δράση μας λοιπόν είναι, όπως είπε και ο διπλανός μου, πρώτα απ' όλα να προσφέρουμε κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες στον κόσμο, στους Λιβύους δηλαδή και κυρίως στους νέους. για να αποφύγουν να αναλάβουν αυτό το καταστραφικό ταξίδι. Επίσης ε, προσφέρουμε και βασικές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της ενέργειας, νερό, κάτι από το οποίο έχουν αποφεληθούν τόσο οι Λίβοι όσο και οι μετανάστες. Η δράση αυτή επίσης θα παραταθεί και θα συμπληρωθεί με μαζική δράση εφόσον έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια και θα συνεχίσουμε από κοινού μαζί με την Ιταλία να βοηθούμε τις τοπικές κοινότητες στη Λιβύη για την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Και τέλος πράγματι θα βοηθήσουμε και τους Λίβιους ακτοφύλακες να γίνουν πιο επαγγελματίε. Η διαδρομή της Μεσογείου, αυτή η μεταναστευτική από την Κεντρική Μεσόγειο, σήμερα είναι η πιο θανατηφόρα. Από το 2015 πάνω από 10.000 άνθρωποι πνίγηκαν στη θάλασσα αυτή. Μειώνεται βέβαια το νούμερο σημαντικά φέτος. Και χωρίς βέβαια να λάβουμε υπόψη μας όλους τους θανάτους που δεν μπορούμε, δεν είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε, που έχουμε στην έρημο της Σαχάρας. Άρα λοιπόν χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία να αποφεύγονται οι αναχωρήσεις πρώτα απ' όλα με αυτό που λέμε σκάφη, αλλά τι σκάφη στην πραγματικότητα είναι αντικείμενα τα οποία κάθε άλλο παραφτιαγμένα για να διασχίζουν τέτοιες θάλασσες είναι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να στηρίζουμε αυτή τη δράση και το 2018 στο δεύτερο στάδιο που θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία μεταξύ άλλων ενός ε, επιχειρησιακού κέντρου για τη διάσωση στη θάλασσα. Αυτή είναι με δυο λόγια η κατάσταση σήμερα όσον αφορά το δικό μας έργο. Τι κάνουμε φέτος και τι θα κάνουμε για τον χρόνο. Ήμουνα λοιπόν σύντομος, ε, τα είπα συνοπτικά και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ο Πρόεδρος Μωράς, ευχαριστώ. Το εκτιμώ αυτό διότι θα υπάρξουν και ερωτήσεις και ήθελα να έχουμε χρόνο για να τις συζητήσουμε. Αυτά λοιπόν από Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, ο Πικέ, επικεφαλής του αρμοδίου τμήματος. Ευχαριστώ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Λίγα λόγια από εμένα εκπρόσωπο της, Επιτροπ... της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Βασικό μήνυμα είναι ότι η ύπατη εκπρόσωπος, κύριε Μογκερίνη, αποδίδει την μέγιστη δυνατή προτεραιότητα στα προβλήματα που θέτει η παράτυπη μετανάστευση στη Λιβύη. Πρώτη στη προτεραιότητα, την οποία μεταφράζει η ύπατη εκπρόσωπος σε διάφορες δράσεις. Πρώτα βέβαια, στον διάλογο που διεξάγει με τους Λίβιους ομολόγους της, αλλά και για άλλα θέματα μετανάστευσης και για τη συνεργασία με τις λιβικές αρχές σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί ανθρώπινη μεταχείριση παράτυπων μεταναστών και προσφύγων και να προχωρήσουν σε συνεργασία οι λιβικές αρχές με τις χώρες μέλη της Ένωσης, βεβαίως, πρωτίστως στην Ιταλία. Το θέμα αυτό ε, είναι συνεχώς το θεματολόγιο της ε, κυρίας Μογκερίνη. Συναντάται με τους ε, ανώτατους αξιωματούχους ε, της ε, Λιβύης αλλά και με εκπροσώπους γειτονικών χωρών ιδίως προς νότον της χώρες Σαχέλ και έχουμε και μια σημαντική βέβαια ε, συνεργασία που πρέπει να οικοδομηθεί με τις χώρες αυτές. Αυτά σε ό,τι αφορά τις πολιτικές δράσεις. Εξάλλου εμείς τις υπηρεσίες εξωτερικών δράσεων σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας της Αρμόδια Γενική Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής προωθούμε αυτή την συνολική προσέγγιση για θέματα παράτυπη μετανάστευσης και προσφυγικού. Μια συνολική προσέγγιση που περιλαμβάνει capacity building, building εκπαίδευση των αρμοδίων λιβικών αρχών, περιλαμβάνει την ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων και των θαλασσίων συνόρων και των χερσαίων. Τρίτο, περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης σε ευάλωτους μετανάστες μέσα στη Λιβύη και στα κέντρα υποδοχής ή κράτησης και τέλος συνεργασία με τους οργανισμούς των, τις οργανώσεις μάλλον των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως το IOM, για την στήριξη εθελοντικών επιστροφών των ε, μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους ο όγκος χρηματοδότησης είναι σημαντικός. Η χρηματοδότηση από χώρε μέλη επίσης υψηλή. Η Ιταλία βεβαίως έχει το νούμερο ένα και άλλες χώρες μέλη οι οποίε έχουν συμβάλει στη χρηματοδότηση του Trust Fund για την Αφρική καθώς και οι χώρες μέλη που συμμετέχουν στις δράσεις ΚΕΠΑ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι σημαντικοί μηχανισμοί τους οποίους έχουμε αναπτύξει και η επιχείρηση UNAFORMED, Σοφία, επιχείρηση δηλαδή που έχει αναπτυχθεί στην Μεσόγειο και έχει διασώσει 42.000 άτομα ε, από τα νερά της ε, Βόρειας Λιβικής θάλασσας καθώς και το πρόγραμμα στήριξης της διαχείρισης των συνόρων που παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της αστάθειας στην Λιβύη αρχίζει τώρα να αναπτύσσει ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και capacity building, building ε, εποφελία των λιβικών αρχών. Και θέλω να τονίσω επίσης ότι μέσα στην εκπαίδευση αυτή η πτυχή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του σεβασμού του ανθρωπιστικού δικαίου αποτελεί το ερυθρό νήμα το οποίο διατρέχει όλες τις δράσεις εκπαίδευσης που εκτελούμε πρόσφατες ειδήσει του CNN για σκλαβοπάζαρα στην Λιβύη βεβαίως έχουν οδηγήσει σε απόλυτη καταδίκη από όλους και βεβαίως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια η ύπατη εκπρόσωπος ξεκαθάρισε απολύτως τις απόψεις της μιλώντας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ε, στην ε, διάσκεψη για την Αφρική, της οποίας προέδρευσε ο πρόεδρος Ταγιάννη και την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ενώσεως, τον πρόεδρο Κόντε και με τον προκαθήμενο της Αφρικανικής Επιτροπής, κύριο Μουσά Φάκη. Και εξέδωσαν μάλιστα κοινό ανακοινοθέν. Με, έχει συζητήσει και με τον πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης IOM για να αναζητήσουν άλλες δυνατότητες σε συνεργασία με τον IOM για να ελαφρύνουν τα δεινά τα οποία υφίστανται οι μετανάστες εντός Λιβύης. Η δράση από τη λιβική πλευρά είναι επίσης αξιοσημείωτη διότι για πρώτη φορά οι λιβικές αρχές εξέδωσαν απόλυτα σαφές ανακοινωθέν που εκφράζει με σαφή τρόπο το γεγονός ότι πρόκειται για κοινή ευθύνη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης, με σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών μέσα στην ίδια την επικράτεια της Λιβύης και βλέπουμε μια αλλαγή στάσεως μέσα στη συζήτηση αυτή και μια προσπάθεια Καθιέρωση μιας καλύτερης συνεργασίας. Ένα θετικό στοιχείο ίσως είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη οι λιβικές αρχές δέχτηκαν μια ομάδα εργασία συντονισμού με συμμετοχή όλων των οργανισμών, των οργανώσεων των ΗΠΑ και βεβαίως και με συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλος παράγοντας που αξίζει να σημειωθεί είναι οι αντιδράσεις αφρικανικών χωρών από τις οποίες ορισμένες τοποθετήθηκαν με πολύ επικριτικό τρόπο απέναντι στην μεταχείριση των προσφύγων και παράτυπων μεταναστών από την λιβική πλευρά, μεταχείριση που στερείται του ανθρωπιστικού στοιχείου, αντέδρασε ευαίσθητα η λιβική πλευρά και για το λόγο αυτό πρόθεσής μας είναι να με την ευκαιρία της διάσκεψης που διεξάγεται σήμερα και αύριο μεταξύ Αφρικανικής Ενώσεως και Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε επίπεδο κυβερνήσεων στο Αμπιτζάν να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την ευκαιρία της διάσκεψης αυτής για να προωθήσουμε περαιτέρω συνεργασία μεταξύ ημών και των Αφρικανικών χωρών που είναι συχνά οι χώρες προέλευσης των προσώπων αυτών και βεβαίω και με συνεργασία της Λιβύης. Και ο ιδιαίτερος στόχος που έχουμε θέσει είναι να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τους αριθμούς μεταναστών που επαναπατρίζονται στις ε, πατρίδες τους σε οικειοθελή βάση. Τέλος και μια προειδοποίηση. Παρά τις ευκαιρίες που βλέπουμε και τις οποίες θα επιδιώξουμε να εκμεταλλευτούμε θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σχετικά με το γεγονός ότι η Λιβύη Βεβαίως παραμένει μια ασταθέστατη χώρα, δεν διαθέτει τους κυβερνητικούς θεσμούς που θα επιτρέψουν στην χώρα αυτή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με αποτελεσματικό και πλήρη τρόπο. Και η παρατήρηση αυτή σημαίνει επίσης ότι η ικανότητα και της Λιβύης και η δική μας να εμπλακούμε σε συνεργασία είναι περιορισμένη. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να επεκτείνουμε την ικανότητα αυτής της συνεργασίας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εν μια νυχτή. Και ως τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να πω ότι βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της παράτυπης μετανάστευση κατά μέτωπον, αλλά θα πρέπει να μην παραμελούμε επίσης το γεγονός ότι μόνη διαρκής λύση για τα προβλήματα της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης και για την ανθρωπιστική μεταχείριση των προσφύγων είναι να επιτευχθεί σταθεροποίηση του λιβικού καθεστώτος και να καθιδηθεί ειρήνη και ασφάλεια στην χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε και τελικά θα ακούσουμε την άποψη της Εστονικής Προεδρίας του κυρίου Μέρτε. Χίτμαν περίπου για 6 λεπτά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που προσκαλέσατε και την Προεδρία και με μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσουμε και τη δική μας άποψη. Θα είμαι σύντομος και θα κρατηθώ σε γενικές γραμμές, γιατί νομίζω ότι οι προελίσσαντες αναφέρθηκαν με αρκετές λεπτομέρειες στο θέμα που συζητάμε. Όταν λοιπόν η κρίση έπληξε και πάλι την Νότια Μεσόγειο τέλη Ιουνίου ε, έφερε την Ιταλία σε δύσκολη θέση ε, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο βάρος εμείς αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Τζάι ε, στις αρχές Ιουλίου και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να συζητηθεί ως βασικό θέμα το ε, πρόβλημα των διαδρομών στη Μεσόγειο. Έπρεπε να παρακολουθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για να διασωθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτό το πρόγραμμα το συζήτησαμε επανειλημμένα τελευταία φορά πριν από τρεις εβδομάδες. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα ε, χρησιμοποιήσαμε και τη στρογγυλή τράπεζα για να εξετάσουμε το θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες αναζητώντας καλύτερες λύσεις. Ο Υπουργός, ο Εστονικός Υπουργός Εσωτερικών και αυτός ε, συμμετείχε ο ίδιος ε, προσωπικά δύο φορές ε, μετέβη στην Ιταλία για να συζητήσει το θέμα με τον Ιταλό ομολογό του. Επισκέφτηκε την Ιταλία επίσης για να συναντηθεί με τους δημάρχους της Ιταλίας τελικά αυτοί δεν ήρθαν όμως τουλάχιστον είχε την πρόθεση. Εξάλλου συμμετείχαμε και στην ομάδα επαφής που ανέφερε προηγουμένως και ο συνάδελφος ε, στην Τίνιδα τον Ιούλιο συνεδρίασε αυτή η ομάδα και τον Νοέμβρη η συνάντηση έγινε στη Βέρνη. Εμείς δεν ήμασταν πολύ κοντά ε, γεωγραφικά σε αυτές τις πόλεις αλλά παρόλα αυτά συμμετείχαμε σε αυτές τις συνεδριάσεις. για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα του προγράμματος είναι απαραίτητο να έχουμε και επαρκή χρηματοδότηση. Αυτό είναι κάτι που το πρεσβεύουν όλα τα κράτη-μέλη. Ε, το θέμα του καταπιστευματικού. Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής και κυρίως ε, το Αφρικανικό παράθυρο που ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος αυτά εδώ και μήνες συζητούνται, συζητήθηκαν στο Συμβούλιο επίσης και τον Οκτώβριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, Υπάρχει λοιπόν ευρεία συνένεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε την υποστήριξή μας προς τη Λιβύη, να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Όσον αφορά στις ε, προτεραιότητες ε, που πρέπει να ε, χρηματοδοτούνται, τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων στα διάφορα κέντρα κράτησης, να βελτιωθούν κοινωνικο-οικονομικά οι κοινότητες στις οποίες βρίσκονται οι μετανάστες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Οκτωβρίου κάλεσε τα κρατη να αναζητήσουν ε, ικανοποιητικούς ε, πόρους και η Προεδρία προσπάθησε να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα συζητήθηκε σε επίπεδο κορεπέρ, στο επίπεδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και επίσης βρίσκεται και στη μερίσια διάταξη των μόνιμων εκπροσώπων. Νομίζω σε αυτή τη φάση μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι και να προσβλέπουμε στην επόμενη χρονιά να υπάρξουν επαρκή κορδίλια για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτό το αφρικανικό παράθυρο για την επόμενη χρονιά. Αυτά είχα να πω προς το παρόν στη διάθεσή σας για εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ερωτήσεις. Τρία λεπτά το πολύ ο καθένας. Γιατί εννοείται όλοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Οπότε αρχίζουμε με την Μπάρμπαρα Σπινέλη. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές και θέλω να πω ότι πραγματικά εκπλήσωμαι από τη διάσταση απόψε που υπάρχει. Μερικοί είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την ανθρωπιστική βοήθεια, από την έκκληση προς τα ενωμένα Έθνη να επεμβαίνουν περισσότερο και πριν από λίγες μέρες ε, υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, με βάση όμως αυτές τις δηλώσεις ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να απαλύρουν τον πόνο των μεταναστών. Υπάρχει λοιπόν διάσταση απόψεων. Και είδαμε όλοι μας το βίντεο του CNN της 12 Νοεμβρίου όπου οι μετανάστες πολλούνται ως σκλάβοι. Αυτά μας τα ξέραμε ευθύς εξ αρχής. Τα ξέρετε. εσείς τα ξέρετε και παρόλα αυτά υπογράψατε συμφωνία με τη Λιβύη. Το 2017 είχε όμως υπάρξει μια συμφωνία όπου αναφερόταν ότι η Λιβύη δεν ήταν ασφαλής χώρα. Τον Απρίλη στα Ηνωμένα Έθνη υπήρξε μια έκθεση σχετικά με την πώληση των μεταναστών ως σκλάβων και υπήρξαν και διάφορες ενώσεις που και αυτές ανέφεραν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν προσφέρεται η απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική βοήθεια στους μετανάστες που κρατούνται στα κέντρα κράτησης. Ε, πρόβλημα είναι και οι συνθήκες διαβίωσης στη Λιβύη που αυτή τη στιγμή είναι μια ε, χώρα πολιτικά παντελώς ανεξέλεγκτη. Αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο κύριος Νομάρχης. Από το 16 μέχρι το 17, από το Μάιο, που εκδιώχτηκαν, αρνηθήκαμε την άφηξη μεταναστών. Αυτό νομίζω το είπατε κι εσείς κύριε Μορκόνε. Έχω λοιπόν μπροστά μου ένα έγγραφο το οποίο πήρα από το Υπουργείο Ιστορικών της Ιταλίας και εκεί αναφέρεται ότι ο αριθμός των ε, ε, εκδιώξεων ε, ή των ατόμων αν θέλετε που δεν δεχθήκαμε από το Μάιο του 16 μέχρι το 17 είναι ο, αυτός που αναφέρεται στο έγγραφο άρα δηλαδή τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι υπήρξε αυτό το γεγονός είπατε αναφερθήκατε σε αυτά που αναφέρει η ε, διεθνής αλληλεγγύη και οι αρμόδιοι του Συμβουλίου της Ευρώπης και είπατε ότι δεν συμφωνείτε με όλα αυτά, με αυτές τις ανοησίες. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτά αναφέρονται σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς από τον προηγούμενο Δεκέμβρη. Άρα νομίζω ότι κάποια στιγμή η Ιταλική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζει την Ιταλική κυβέρνηση θα πρέπει να σχίσουν, να κατανοούν ότι αυτές οι ανοησίες δεν είναι απλά ανοησίες, είναι πραγματικότητα. Πρόεδρος. Όντω, ε, ναι, καλείστε να απαντήσετε, αλλά παρακαλώ κάντε λίγο υπομονή να ακούσουμε και τις άλλες ερωτήσεις. Θα σας δώσω το λόγο στο τέλος. Ακόμα και αν είναι προσωπικές κάποιες παρεμβάσει που ακούμε. Ε, παρακαλώ, κύριε Σλάιν. Σας ε, καλωσορίζουμε και πάλι, κύριε Νομάρχα η μεταρρύθμιση της συμφωνίας ε, του Δουβλίνου ε, που προβλέπει και την ε, ευθύνη των κρατών μελών για το θέμα της υποδοχής. Αυτό είναι η δική μας η προσπάθεια, αλλά φοβάμαι ότι αυτά δεν βρίσκουν απήχηση. Γιατί δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να θεωρεί ότι το πρόβλημα πρέπει να μετατεθεί στο εξωτερικό. αλλά για να λυθεί ένα πρόβλημα δεν είναι το να το αγνοεί κανείς απλώς. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει υπάρχει ε, καθυστέρηση. Τέσσερι ώρε αναφέρθηκε ότι υπήρξε την τελευταία φορά. Πέθαναν πολλοί άνθρωποι και ένα μωρό, ενώ οι ε, λιβικές αρχές ε, που υποστηρίχτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' ουσίαν καθυστέρησαν ε, και ε, παρεμπόδισαν και την παρέμβαση της Sea-Watch οι Λίβοι κατ' ουσίαν ε, δεν βοήθησαν καθόλου τους ε, μετανάστες οι οποίοι ε, βούτυξαν στη θάλασσα και δεν άκουσαν καθόλου και τις αγωνίες, κραυγές αγωνίες που είχαν εκφράσει οι Ιταλοί. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στην Λιβύη. Βλέπετε ότι συνεχίζεται η ίδια εγκληματική συμπεριφορά παραβιάζονται οι διατάξεις περί επαναπροωθήσεων. Υπάρχει λοιπόν μια, ένα κενό στην Μεσόγειο και ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια μεγαλύτερη προσπάθεια για να εφαρμόζονται οι θεσμικές διατάξεις ε, σχετικά με τη διάσωση των ζώων στη θάλασσα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας αποτελεσματικός έλεγχος. Ε, ο ύπατος εκπρόσωπος, ύπατη εκπρόσωπος για τους πρόσφυγες αναφέρει ότι αυτά τα οποία έγινε στη Λιβύη κατ' ουσίαν τα, ξέραν, τα ήξεραν όλοι. Το Associated Press αναφέρει ότι τελικά τα χρήματα που οποία δίδονται υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουν ε, στους λαθροδιακινητές. Ο μόνος ε, τρόπος ε, για να αντιμετωπιστούν οι λαθροδιακινητές είναι όχι να τους πληρώνουμε αλλά να ανοίξουμε τους, τις οδούς για να μπορούν να έρχονται μετανάστες. Μπορούν να γίνουν συγκρίσεις αριθμών και θα καταλάβουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές ε, υπό, την, ε, υπό τον έλεγχο των λιβικών αρχών. Θέλω να πω το 10 εκατομμύρια έχει δώσει η Ιταλία ε, και άλλα 42 εκατομμύρια για το καταπιστευματικό ταμείο για να ελέγχονται τα σύνορα στην Λιβύη. Η Ιταλία θεωρεί ότι πρέπει να προωθήσει τα δικά της τα συμφέροντα το 90% των κονδυλίων προέρχονται όμως από κονδύλια για την ανάπτυξη που αυτή τη στιγμή ακολουθούν τελείως διαφορετική πορεία που δεν είναι όμως με βάση το συγκεκριμένο άνθρωπο που προβέται στη συνθήκη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το Υπουργείο Εστερικών εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να το ελέγχει. Θέλουμε να έχουμε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα για το πώς ακριβώς γίνονται οι δαπάνες. Η ε, Κομισιόν απάντησε σε μια δική μας ερώτηση αλλά ήταν ε, πολύ αφηρημένη η απάντησή της και λέει ότι ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται από την Ιταλία και από τρίτους και θα θέλαμε να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι τρίτοι οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν αυτόν τον έλεγχο. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη. Ε, δεν σας προλάβαινα. Είπαμε τρία λεπτά ο καθένας. Και να μιλάτε και λίγο πιο αργά. Ακόμα και αν έχετε να πείτε πολλά, ε, δεν πρέπει να τρέχετε έτσι, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Λάρα. Όχι όμως πολύ γρήγορα, έτσι σε παρακαλώ. Πριν από λίγες μόνο εβδομάδες η συμφωνία ανάμεσα στην Ιταλία και τη Λιβύη χαρακτηρίστηκε απάνθρωπη αυτή η συμφωνία από τον αρμόδιο επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ράπισμα για την ε, ανθρωπιστική στάση γιατί γίνεται λόγος ε, για αυθαίρετες κρατήσεις γίνεται λόγος για βασανιστήρια για βιασμούς για εκβιασμούς το CNN έδειξε ότι στη Λιβύη υπάρχει παζάρι με μετανάστες που πολλούνται ως δούλοι στην Ιταλική τηλεόραση είδαμε ένα βίντεο όπου βλέπουμε αστυνομικούς ε, της ακτοφυλακής ε, της Λιβύης που χτυπάνε τους ε, μετανάστες. Μερικοί έχουν πιαστεί από το σκάφος και το Ιταλικό ελικόπτερο προσπαθεί να μπλοκάρει όλη αυτή τη διαδικασία. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση προς τον κύριο Μορκόνε. Θα ήθελα να γνωρίζω αν τελικά για όλα αυτά έχει γίνει κάποια έρευνα, γιατί εδώ πρόκειται για κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, οι Λίβοι ε, παίρνουν τα χρήματά μας αλλά δεν γίνεται κανένας έλεγχος επί τόπου. Ο έλεγχος γίνεται άμεσα ή έμεσα από ομάδες ε, οι οποίες ε, διαχειρίζονται την διακίνηση των ε, μεταναστών. Και από εκεί εξαρτάται πόσοι θα έρθουν στην Ιταλία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να κάνω τις εξής ερωτήσεις. Γιατί δεν υπάρχει μία αναγνωρισμένη αρχή στη Λιβύη με την οποία να μπορούμε να συζητήσουμε. Όταν μιλάμε για τη Λιβική ακτοφυλακή θα ήθελα να γνωρίζω ποιους ακριβώς πληρώνουν κάνουμε. Ποια είναι, ποια, είναι, είναι εκείνη η περιοχή στη Λιβύη που ελέγχεται και από ποιον. Στη Λιβύη η Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά κάνουν πόλεμο κατά των διακινητών ή κατά των μεταναστών. Αυτό δηλαδή που μας ενδιαφέρει είναι να μην έρθουν σε εμά μετανάστες με οποιοδήποτε τίμημα και ποιος ελέγχει τα κέντρα κράτησης ε, στη Λιβύη και αυτά τα κέντρα παίρνουν χρήματα από την Ιταλία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα παρακαλώ να μου απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους πάρα πολλές ερωτήσεις θα σας δώσω αρκετό χρόνο για να απαντήσετε Η Κατερίνα Κινίτση έχει τώρα το λόγο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, καλεσμένους μας. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν παρούσα από την αρχή, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Νομάρχης ε, σας εξήγησε το τι ακριβώς κάνει η Ιταλία για να υποδέχεται τους ε, μετανάστες και να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση στην επικράτειά μας. Βεβαίως κάποιες ερωτήσεις δικές μου ήδη ετέθησαν, δηλαδή η Ιταλία έχει συνάψει κάποιες συμφωνίες με τη Λιβύη, αλλά με τον τρόπο αυτό δεν απεκδίεται των ευθυνών της. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων ε, που βρίσκονται σε κέντρα κράτηση στη Λιβύη. Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι συνθήκες είναι δραματικές και αναφέρομαι κυρίως στους ανήλικους ε, για τους οποίους πιστεύω ότι ποτέ δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται η κράτησή τους. Απλά και μόνο για το γεγονός ότι είναι ανήλικοι και μετανάστες. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Έχουν γίνει κάποια, αλλά ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά. Να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες, να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα παρότι ο ύπατος εκπρόσωπος για τους πρόσφυγες έχει επισκεφτεί αυτά τα κέντρα. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι το συντομότερο δυνατόν να γίνεται έλεγχος ε, για το ποιοι ακριβώς ε, διαχειρίζονται τα κέντρα αυτά, κυρίως όσον αφορά τους, ε, τις πιο ευάλωτες περιπτώσεις. Στην περίπτωση των οικειοθελών επιστροφών, αυτό να γίνεται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα ήθελα να ρωτήσω και πολλά άλλα πράγματα, αλλά τα έχουν ήδη ερωτήσει οι προελίσσαντες. Και θα μου επιτρέπετε να πω το εξή. Το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω. Κατά τη δική μου άποψη δεν έχει εξευρεθεί ακόμα η ε, σωστή αντιμετώπιση της λαθροδιακίνησης γιατί εξακολουθεί να υπάρχει η λαθροδιακίνηση παρά τις διάφορες παραμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν οι λάθροδιακινητές και αν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα θεωρώ ότι θα συνεχίσει να υπάρχει παραβίαση και κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα όχι ως μεμονωμένη χώρα, ως Ιταλία, να το αντιμετωπίσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Να καθορίσουμε τις ευθύνες που πρέπει να, να αναλάβει ο καθένα. Αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, θα συνεχίσει να υπάρχει λαθροδιακίνηση και δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τίποτα. Ευχαριστούμε, η Μαλίν Μπιόρκ. Ευχαριστώ πολύ. Οφείλω να πω ότι ανησυχούσα πριν και τώρα ακόμα περισσότερο, έχοντας ακούσει τους προσκεκλημένους μας. Η κατάσταση, όπως υπογραμμίζουν οι συνάδελφοι, είναι πέρα από αυτά που θα μπορούσε να αντέξει κανείς να δει. Εντάξει, υπάρχει το κρατός δικαίου, η δημοκρατία, η λειτουργία της κοινωνίας, όλα αυτά αναφέρονται, ναι. Οπότε ρωτάω, ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Λιβύη. Το λέω αυτό για το Σεβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τι είναι η καταπολέμηση της παράτυπης ε, Μετανάστευση αυτό είναι όλο. Δεν πρέπει να δούμε μήπως είμαστε και εμείς τελικά ε, στη Λιβύη για παράδειγμα μέρος του προβλήματος. Και έπειτα, σήμερα το πρωί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κρόαση και κάποιοι πυρογνώμονες είπαν ότι οι περισσότεροι που επιστρέφουν, επιστρέφουν καταναγκαστικά και κάτω από πολύ κακές συνθήκες. Ποιος τα ελέγχει όμως όλα αυτά δεν έχουμε καμία εγγύηση για τους ε, εταίρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Η Λιβική ακτοφυλακή λειτουργεί με έναν τρόπο παράδεκτο, το ξέρουμε, τους, ε, έχει τους ανθρώπους κάτω από απέσχες συνθήκες, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να εμποδίσουμε τους ε, Λίβιους να το κάνουν αυτό, να μην γυρνάνε οι άνθρωποι στις φυλακές. Αυτά για να ξέρουμε ποιους εταίρους υποστηρίζουμε. Και ρωτάω λοιπόν, ποιοι είναι στα ε, νότια σύνορά μας οι εταίροι μας, ποιοι είναι αυτοί που είναι ε, οι αποδέκτες της οικονομικής μας βοήθειας. Και η τρίτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τους καταβλισμούς κράτησης. Κανένας από αυτούς τους καταβλισμούς δεν είναι σε αποδεκτή κατάσταση πώς να τα εξηγήσω όλα αυτά στους ψηφοφόρους μας. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση εκεί. Εμείς πρέπει να ζητήσουμε να κλείσουν αυτοί οι κατευλισμοί. όχι να τους διατηρούμε ανοιχτού. Και όσον αφορά τις επιστροφές. Όταν μιλάτε για επιστροφές σε εθελοντική βάση, ε, αυτό ακούγεται πολύ περίεργο. Όταν κάποιος είναι κάπου κλειδωμένος, ε, τι επιλογή του δίνεται. Δεν είναι σωστή αυτή η διατύπωση, τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση της Λιβύης. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κώστερ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Κώστερ. Κύριε Πρόεδρε, είχα ήδη από την αρχή την εντύπωση ότι η κατάσταση στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβύης εμφανίζεται κάπως ωρεοποιημένη. Νομίζω ότι η κατάσταση θα πρέπει να περιγραφεί με τρόπο ρεαλιστικότερο, όπως το έκαναν μόλις πριν οι ε, συναδελφοί μου που μίλησαν πριν από μένα. Έχω το εξή παράδειγμα που δείχνει τη δραματικότητα της κατάστασης. Της 6 ενδεκάτου έγινε ένα βαρύ επεισόδιο στην Μεσόγειο, όπου με παρέμβαση της Λιβικής Ακτοφυλακής έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ένα μικρό παιδί. Ένα φουσκωτό με πρόσφυγες είχε στείλει ε, και με υποστήριξη ενός γαλλικού σκάφους και ενός ιταλικού ελικοπτέρου προσπαθούσαν να διασώσουν τους ε, ναυαγούς από τον πνιγμό. Εκτός των 30 μιλίων, ένα σκάφος της Λιβικής Ακτοφυλακής πέραν παντός ορίου δικαίου παρεμπόδισε την ε, παρεμβασία αυτή. Αποτέλεσμα πέθαναν πέντε πρόσφυγες. Εάν η Λιβική Ακτοφυλακή είχε τηρήσει το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, αυτή η καταστροφή θα είχε αποφευθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλαπλές σχέσεις με τη Λιβική ακτοφυλακή. Εκπαίδευση, χρηματοδότηση, παροχή υλικού και επομένως υπάρχει συνευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα πώς αξιολογεί το επεισόδιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ακριβώς κάνει για να ερευνήσει το θέμα αυτό. Και από αυτό απορρέει άλλο ερώτημα. Υπάρχει κάποια ε, συγκεκριμένη εκπαίδευση τη Λιβική Ακτοφυλακή μπορούμε να τη δούμε εμεί ω Ευρωβουλευτέ. Υπάρχει κάποια έκθεση monitoring, παρακολούθηση από ανεξάρτητα όργανα. Η Λιβική Ακτοφυλακή τον τελευταίο καιρό έχει κατ' επανάληψη παραβιάσει το διεθνέ δίκαιο. Και επιτέλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αναλάβει δράση ώστε το διεθνέ δίκαιο να τηρείται στην πράξη και όχι μόνο με λόγια. Εν ώψη της τραγικής αυτής ιστορίας αλλά και πολλών άλλων που συμβαίνουν γύρω από τη Λιβύη είναι απολύτως αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την πολιτική της απέναντι στη Λιβύη και να επανέλθει μέσα στο πλαίσιο τήρησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τους ε, ομιλητές για τις προφορίες που παρέσχουν. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ασαφή για μένα. Και σκέπτομαι αυτό που είπατε για την προτεραιότητα. Ότι η προτεραιότητα είναι η δίωξη των λαθροδιακινητών. Σαφώς συμβαίνει αυτό. Αλλά διαρωτώ με τι μπορεί να κάνει κανείς στην περίπτωση αυτή όταν αντιμετωπίζει λαθροδιακινητές στα σκάφια αυτά. Πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν στην Ιταλία. Θα αφήσετε λοιπόν να μετακινηθεί το πρόβλημα εκεί. Μιλούμε τώρα για σκάφη που κινούνται κοντά στις λιβικές ακτές. Τι γίνεται, προσπαθούν να μεταφέρουν τους ε, πρόσφυγες ξανά στη Λιβύη, τους αφήνουν να πάνε στην Ιταλία. Τι ακριβώς γίνεται. ρωτώ με επίσης, μιλήσατε για μείωση 32% των μετακινήσεων από τη Λιβύη προς την Ιταλία. Ίσως αυτό που βλέπουμε όμως για παράδειγμα σε άλλες χώρες όπου η Ισπανία βλέπουμε αύξηση των αφήξεων έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των προσώπων που φτάνουν στην Ισπανία από πέρσι 500.000 έχουν φτάσει οι παρατημετανάστες στη Νότια Ισπανία έχουμε από τη μια μεριά τη συμφωνία με την Τουρκία που δεν αποδίδει και είναι ζήτημα χρόνου μέχρι να αρχίσουν να μας ζητούν περισσότερα χρήματα. Αυξάνουν οι αριθμοί των αφήξεων στην Ελλάδα ούτως ή άλλως. Μετά έχουμε τη Λιβύη. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Θα διαπραγματευτούμε με το Μαρόκο. Νομίζω ότι ο πιο ανθρωπιστικός τρόπος είναι να πούμε όχι. Η Ευρώπη έκανε το καθήκον της. Κάθε κυβέρνηση φροντίζει τα της χώρας της. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε ένα στόπ σε όλους αυτούς τους θανάτους στη Μεσόγειο, λέγοντας απλώς όχι. Τις τελευταίες ημέρες ε, πήραμε πάρα πολλές ε, ειδήσει σχετικά με το σκλαβοπάζαρο στη Λιβύη. Αυτό απλά επιβεβαιώνει αυτό το οποίο γνωρίζαμε εδώ και πολύ καιρό. Ε, πολλοί από τους εκλογεί μου, τους δικούς μου τουλάχιστον, με ρώτησαν τελικά τι συμβαίνει. Είχαν, ήταν συγκλονισμένοι άνθρωποι και εγώ είμαι εξοργισμένο ε, που δεν άκουσα σήμερα τίποτα για το συγκεκριμένο γεγονός. Ε, ε, το αποφύγατε και είμαι και ε, ξοργισμένος για την αδυναμία που επιδείξατε. Σαν δηλαδή να είναι κάτι που απλά το δεχόμαστε. Αν θέλει κανείς να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη λαθροδιακίνηση και όλα τα άλλα φοβερά συμπαρομαρτούντα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το, τη λαθροδιακίνηση δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με τους ε, αυτή είναι μια ολέτρια αντιμετώπιση του προβλήματος που κατ' ουσίαν εκφράζει μόνο την αδυναμία. Εμένα θα με ενδιαφέρε το κατά πόσον μπορείτε να μας αναφέρετε συγκεκριμένους αριθμούς. Για πόσους ανθρώπους ε, μιλάμε, πώς είναι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στη Λιβύη, γιατί ε, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και φοβάμαι ότι δεν έχετε καν συγκεκριμένους αριθμούς. Για πόσους ανθρώπους τελικά μιλάμε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λούζιν είναι η επόμενη μιλήτρια. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ πρέπει να σας πω ότι πραγματικά έχω τρομάξει με αυτά τα οποία άκουσα. Αλλά κυρίως έχω τρομάξει με αυτά τα οποία δεν υπόθηκαν. Και έχω τρομάξει και με την μονόπλευρη θεώρηση των πραγμάτων που αφορούν στη Λιβύη και κυρίως τα ύδατα μπροστά από τη χώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα με εκπροσώπους ε, της Sea-Watch ε, και της ε, οργάνωσης Γιατροί χωρι Σύνορα. Εκεί λοιπόν μου αναφέρθηκαν και άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο αυτή την οποία ανέφερε ένας από τους προλαλήσαντες. Είδα λοιπόν συγκεκριμένες εικόνες για το πώς η ακτοφυλακή κατέστρεψε ένα φουσκωτό, το έσκησε με μαχαίρια. Οι άνθρωποι της Sea-Watch ήθελαν να σώσουν τους μετανάστες που βρισκόντουσαν στο φουσκωτό και ξέρετε τι έγινε. Οι άντρες της ακτοφυλακής απείλησαν τους ανθρώπους με όπλα και τους ε, εμπόδισαν και τους ανθρώπους της Sea-Watch να σώσουν τους άλλους που είχαν πέσει μέσα στη θάλασσα. Ε, πίσω στο βάθος έβλεπε κανείς και άλλα σκάφη. Τώρα δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν σκάφη της ε, Ιταλικής ακτοφυλακής. Πάντως υπήρχαν κάποια σκάφη τα οποία απλά παρακολουθούσαν. Δεν έκαναν τίποτα. Παρακολουθούσαν την κατάσταση. Αυτά ξέρετε δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα. Οι άνθρωποι από τους γιατρούς χωρίς ώρα και από τη Sea-Watch μου είπαν ότι αυτό ε, διαδραματίζεται σχεδόν κάθε μέρα. Και δεν είναι δυνατόν τόσο οι Ιταλικές αρχές όσο και οι Λιβικές ε, οργανώσεις να μην τα γνωρίζουν όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν. Όλα αυτά γίνονται υπό την αποδοχή, γίνονται στα μάτια όσων παρίστανται και γι' αυτό λοιπόν εγώ πραγματικά ε, συγκλονίζομαι και εγώ που ακούω όλες αυτές τις μεγαλοστομίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και για τα μέτρα διάσωσης. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εδώ δεν πρόκειται για μέτρα διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ακριβώς αυτό το οποίο ανέφερε η συνάδελφος από τη Σουηδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι στους πρόσφυγες και λέει και όχι στην ε, επιβίωση των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται σε ε, φυγή. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω και ποιος είναι ο κώδικας ε, που ισχύει για την εκπαίδευση της ε, λιβικής ακτοφυλακής και ποιες είναι οι νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν. Και έχω και μία ερώτηση προς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το οποίο αναφέρεται ως βιώσιμη λύση. Αυτό το βιώσιμη λύση τελικά Πώς ακριβώς το εννοείτε, κυρίως έχοντας κατά νου ότι εντωμεταξύ ε, πεθαίνουν στην έρημο τρεις φορές περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι στη Μεσόγειο. Δηλαδή αυτό τώρα τι είναι, είναι βιώσιμο το να λέμε ότι πυροβολούμε τους ε, ανθρώπους ε, στη θάλασσα ε, για να μην αναγκαστούν να ξανάρθουν μέσω θαλάσσης και να πηγαίνουν μέσω ερήμου και εκεί όμως βλέπετε ότι και αυτοί τελικά καταλήγουν δεν είναι η λύση το να γύρουμε όλο και περισσότερα τείχη και σύνορα. Ε, εσείς δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να επιδείξετε μια πιο ανθρωπιστική στάση όσον αφορά την βιώσιμη ανθρωπιστική πολιτική. Ο κύριος Κόρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ε, θα είμαι ε, πάρα πολύ ε, σύντομος. Ε, ελέγχθησαν πάρα πολλά από τους ε, συναντέλφου και υπάρχουν ε, δύο πράγματα που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Νομάρχη. Το πρώτο πράγμα αφορά τα χρήματα. Θα ήθελα να κατανοήσω κατά πόσον σε αυτή την επιχείρηση με τη Λιβύη σε τελική ανάλυση η Ιταλία είναι εκείνη η οποία εκταμιεύει τα κονδύλια ή αν θέλετε τελικά πόσα χρήματα έχουν διατεθεί για αυτές τις επιχειρήσεις. Και όσον αφορά αυτό το καταπιστευματικό ταμείο, ξέρετε αυτό κατ' ουσίαν θα έπρεπε να έχει ως στόχο την ανάπτυξη και όχι τον έλεγχο των συνόρων. Θέλω λοιπόν να γνωρίζω ε, τι γίνεται και σε περιπτώσεις άλλων συμφωνιών, γιατί υπάρχει και συμφωνία με την Τουρκία, παραδείγματο χάρη. Θα ήθελα να γνωρίζω αν η Ιταλία για άλλη μια φορά έχει αφαιθεί μόνη τη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και οικονομικά. Και αυτή ήταν η μία ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι κατά πόσον ε, βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια λύση. Ε, εσείς ε, έχετε συνεργαστεί στενά με τον Υπουργό, θα έχετε ακούσει για τα βασανιστήρια, για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ε, το Υπουργείο πώς ακριβώς αντιμετωπίζει την κατάσταση. Η Ιταλία έχει σκεφτεί κάποιες λύσεις και θα ήθελα να ξέρω και κατά πόσον σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια ερώτηση και προς τους άλλους τρεις καλεσμένους. Ε, σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρίξει φως ε, σε όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται στη Λιβύη. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κ. Τσέζη. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές. Κυρίως ε, τον Νομάρχη κύριο Μορκόνε. Να τον ευχαριστήσω ως Ιταλός εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στην αντιπολίτευση, αλλά παρόλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας ε, τον Υπουργό Ιστερικών ε, της χώρας μου, που τον τελευταίο καιρό κάνει καταπληκτική δουλειά. Καταπληκτική δουλειά στη Λιβύη. Μάλιστα έκανε και συνάντηση με τους δημάρχους των παράκτιων κοινοτήτων και περιοχών Πολλές ερωτήσεις ε, έχουν ήδη τεθεί από τους προλήσαντες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ουσιαστικό θέμα. Τι κάνει τελικά η Ευρώπη. Εντάξει, η Ιταλία ήδη κάνει πάρα πολλά. Εμείς ε, οι Ευρωπαίοι και αυτοί που είμαστε εδώ, οι Ευρωβουλευτές, πώς βοηθάμε την Ιταλία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Το πρόβλημα κατ' ουσίαν είναι τι κάνουμε για να σταθεροποιηθεί η Λιβύη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ιταλία να κάνει μόνη της όλη αυτή τη δουλειά. Άρα αυτή την ερώτηση δεν την απευθύνω ε, μόνο στον κύριο Μερκόνο, αλλά γενικότερα τι κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι, τι κάνει το Συμβούλιο και η Κομισιόν για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Λιβύη. Γιατί αν δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Λιβύη, απλά ξέρετε κάτι, θα λέμε ωραία λόγια και τίποτα παραπάνω. Σας το λέει κάποιος που είναι στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, ο υποφαινόμενος. Γι' αυτό λοιπόν Θέλω να ερωτήσω τους ε, παριστάμενους, γιατί έχουμε εκπρόσωπο και της κυρίας Μογκερίνη και του Συμβουλίου, να μας πείτε τι κάνετε για να σταθεροποιήσετε τη Λιβύη. Αν δεν σταθεροποιηθεί η Λιβύη, κατ' ουσίαν σας λέω, απλά συζητάμε χωρίς συγκεκριμένο λόγο άνευ ουσίας γιατί ε, ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές και δεν θα κατορθώσουμε ποτέ να αναχαιτήσουμε την έξοδό τους. Τελικά γιατί πράγμα ακριβώ συζητάμε. Δεν μπορούμε να αναθέσουμε αυτή τη δουλειά μόνο στην Ιταλία. Σας το λέω ως Ιταλός, ε, αυτά τα οποία σημαίνουν είναι απαράδεκτα, γι' αυτό λοιπόν εγώ ερωτώ τους εκπροσώπους ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του Συμβουλίου τι κάνετε. Τι κάνετε για να προκύψει μια πολιτική λύση στη Λιβύη, γιατί αλλιώς σας λέω απλά θα συνεχίσουμε να συζητάμε ανεπλογού και briefly. Τελευταίος ήταν τελειώσει το τηλέφωνό του. Παρακαλώ Τόμας, κύριο Ζητερνόφσκι. Ε, ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν επιθυμώ να επικρίνω την Ιταλία, διότι πιστεύω ότι η Ιταλία έχει επιτύχει σε πολλές πτυχές της προσπάθειάς της και χρειάζεται υποστήριξη από όλους μας. Τους πρόσφατους μήνες, εάν η Ιταλική κυβέρνηση δεν είχε κάνει κάποια βήματα, δεν είχε λάβει κάποια μέτρα, ολόκληρη η Ευρώπη θα είχε γεμίσει εξτρεμιστές. Γι' αυτό, αγαπητέ κύριε Μορκόνε, να θέσω μια ερώτηση σχετικά με τη συνεργασία σας με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Συνεχίζω στα αγγλικά. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να σας ευχαριστήσω. Συνεχίστε Τόμα, συνεχίστε. Ευχαριστώ λοιπόν για την θαυμάσια δουλειά που κάνετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Ιταλικούς θεσμούς. Συνεχίστε το μας, ε, λέει ο Πρόεδρος. Ερώτηση λοιπόν. Συνεργασία με μη κρατικές οργανώσεις στη Μεσόγειο, μη κυβερνητικές οργανώσεις στη Μεσόγειο. Πώς διαμορφώνεται η συνεργασία αυτή τώρα. πώς καταφέρνετε να υλοποιήσετε τα όσα είχατε προτείνει ήδη από το καλοκαίρι. Δεύτερο, το μέλλον της συνεργασίας με τις λιβικές δυνάμεις. Πώς βλέπετε να διαμορφώνετε. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα εκεί. Επίσης, οι Ιταλικές ναυτικές δυνάμεις, ε, πώς μπορούν να επιχειρούν σε λιβικά ύδατα και με ποιο τρόπο να ανακόπτουν τα ρεύματα των παρά μεταναστών και προσφύγων. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μολκόνε, διότι του τέθηκαν πολλές ερωτήσεις ευθέω. Πήγε δική μας αντιπροσωπεία τον προηγούμενο μήνα στην Τινησία. Ισία. Είδαμε και εκπροσώπους της Λιβικής Ακτοφυλακής, όπως θα επιβεβαιώσει και η κυρία Βερουζιά. Έγινε μια αποστολή, μια ε, έρευνα από μέρους μας σε βάθος δεν θέλω να υπάρξει καμιά παρανόηση. Πήγαμε εκεί, ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά, γνωρίζουμε ποιε είναι οι περιπλοκέ ε, του θέματο και αντιλαμβανόμαστε το μέγεθο τη ε, προσπάθεια. Είμαι βέβαιος ότι αυτά τα λόγια μου μπορεί να επιβεβαιώσει και η κυρία Βεργία. Παρακαλώ, προσπαθήστε κύριε Μόρκον να απαντήσετε σε όσο γίνεται περισσότερε από τι ερωτήσει που σα τέθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο. Αυτό το είπαν και κάποιοι ευρωβουλευτές. Ε, να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για την πολύ καλή δουλειά που κάνει για τη μεταρρύθμιση, τροποποίηση μάλλον, της Συμφωνίας του Δουβλίνου. Εμείς, ε, η Ιταλία, εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτή την προσπάθεια και ε, προσβλέπουμε και στα αποτελέσματα προσβλέπουμε στο να ευοδοθούν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένδειξη πραγματικής αλληλεγγύης και αναγνώριση του ότι πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες. Ξέρω ότι πρέπει να τα πω γρήγορα, αλλά τι να κάνω, θα τα πω, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Λοιπόν, όσον αφορά τις ΜΚΟ, όλοι υπέγραψαν εκτός από την MSF. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ 44 χρόνια α, ασχολούμαι με τον τομέα, τα τελευταία χρόνια με τη μετανάστευση. Όλοι υπέγραψαν, όλοι είναι επιτόπου και εργάζονται α, ε, χωρίς ε, ουσιαστικό περιορισμό. Όσον αφορά τώρα ε, τη στάση της Ιταλίας. Ε, πράγματι η Ιταλία δεν είναι ε, ικανοποιημένη, δεν θεωρεί ότι υπάρχει απαραίτητη αλληλεγγύη. Σας είπα ότι εγώ από το 2006 ασχολούμαι με τα θέματα των δικαιωμάτων και της μετανάστευσης και σήμερα πάρα πολύ ένας γνωστός Λίβιος που δεν θέλω να προσβάλλω. Όλοι λένε ότι εκπλήσονται, αλλά εγώ τα ξέρω τα πράγματα από το 2006. Η Ιταλία λοιπόν αποφάσισε βλέποντας το ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει σταθεροποίηση της Λιβύης, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα, να υπάρξει δημοκρατική νοοτροπία και πολιτισμός από τη χώρα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Αναγνωρίζοντας η Ιταλία ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η ζωή των ανθρώπων, αποφάσισε να συνάψει μία συμφωνία με τη Λιβύη, η οποία συμφωνία εγκρίθηκε και από τον Αθήνα Δεν εγκρίθηκε από το φίλο μου στον δρόμο, Αποφασίσαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο και αυτό, όπως σας είπα, για να στηρίξουμε όχι μόνο τη Λιβύη, αλλά και άλλες χώρες της Αφρικής. Γιατί κατά την άποψή μας, ένα θέμα που εγκαταλείψαμε εδώ και πολλά χρόνια είναι η ανάπτυξη και τα δικαιώματα και ο σεβασμός των ανθρώπων στην Αφρική. Στη Λιβύη, αλλά και σε άλλες χώρες, και στον Βορρά και στον Νότο. Όχι ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε άλλες χώρες. Και νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ από εσά που έχετε πάει και τα έχετε δει. Κύριε Κώστα, Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ε, συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά πράγματι ε, υπάρχουν σοβαρές ποινικέ καταστάσεις και πράξεις. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει πάση θυσία να αντιμετωπίσουμε τη λαθροδιακίνηση, να καταστρέψουμε τη λαθροδιακίνηση. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε ένα βήμα προς την κατεύθυνση του σεβασμού της ζωής και των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Αυτή είναι μια αρχή προς την οποία μετακινούμε τα εμείς αυτή τη στιγμή ως χώρα, ως Ιταλία. Τώρα, η εκπαίδευση της ακτοφυλακής, της λιβικής ακτοφυλικής. Όπως σας είπα, αυτό είναι ένα θέμα της ίδιας της Λιβύης και η εκπαίδευση γίνεται με βάση ε, διεθνείς προδιαγραφές που όλοι τις γνωρίζετε. Πολύ επικαλείστε τα γεγονότα της 6ης Νοεμβρίου. Και εγώ τα είδα αυτά στην τηλεόραση, όπως επίσης ε, και είδα και στο facebook όπου οι Λίβοι προέβαλαν τη δική τους την ιστορία. Εγώ δεν θέλω να κρίνω αν έχει δίκιο ο ένας ή ο άλλος. Απλά θέλω να πω ότι ε, ξεκίνησε η διαδικαστική διαδικασία του θέματος επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη και πλέον θα αποφανθεί σχετικά με τους κανόνες. Το ίδιο νομίζω ισχύει και για όλες τις άλλες ε, παρατηρήσεις και για όλα τα άλλα σχόλια που αναφέρθηκαν. Ε, θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι ακράδαντα πεπισμένος και είμαι και υπερήφανος ε, για αυτά που έκανε η πατρίδα μου τελευταία χρόνια. 700.000 δεχτήκαμε. Εκτός από την Ιταλία Άλλοι φίλοι μας στην Ευρώπη δεν δέχτηκαν ούτε μία ΜΚΟ. Εμείς δεχτήκαμε 700.000 άτομα. Και κύριε Σπινέλη, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό. Αυτά που λέει η Διεθνής Αμνηστή, όχι μόνο είναι ανοησίες, είναι και λάθος, είναι ψέματα. Αν θέλετε να με καταγγείλετε, εγώ σας λέω, δεν μπορούν αυτά να τα αποδείξουν που λένε ότι χρησιμοποιούν ηλεκτροσόκ. Ίσως να πηγαίνουν πολύ συχνά στο σινεμά οι φίλοι της Διεθνούς Αμνηστίας και να βλέπουν το Ράμπο γιατί ε, δεν υπάρχουν αυτά τα ηλεκτροσόκ στην Ιταλική αστυνομία. Δείξτε μας έστω και μία φορά. Αυτά είναι πολύ γενικά που λέγονται και επαναλαμβάνω. Οι διεθνεί ο αμνηστή, αυτά που λένε είναι ψέματα. Και πρέπει να πω, κυρία Σπινέλη, λυπάμαι πάρα πολύ, σας το λέω. Ε, εσείς ε, Είσαστε πολλά χρόνια ε, στην πολιτική και διαβάζετε πάρα πολλά. Εγώ θέλω να σας πω λοιπόν ότι η Ιταλία ποτέ δεν έδιωξε κανένα. Κανένα μετανάστη που να θέλει να έρθει σε εμάς. Πριν διαβάσετε αυτό που θέλω να μου πείτε, εσείς μιλάτε ε, για ανθρώπους ε, τους οποίους ε, δεν δεχτήκαμε Εντάξει, αυτό που λέει ότι μέσα σε 7 μέρες έχουμε δικαίωμα να τους ε, επιστρέψουμε, αυτό είναι κάτι τελείως ε, διαφορετικό. Η τινήση είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ζητούν άσυλο, μόλις αποβιβαστούν. Μετά αν θέλετε εντάξει να τα δούμε τώρα μαζί αυτά που μου λέτε. Δεν νομίζω ότι αυτά που ε, λέτε ενδιαφέρουν όλους του ευρωβουλευτέ, Μετά να τα δούμε κατηδίαν. Η Ιταλία είναι υπερήφανη για αυτά τα οποία κάνει και θέλω να σας πω ότι με τους φίλους, τους Γερμανούς, τους Γάλλους ε, και από πολλές άλλες ε, ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες ε, συμμετέχουν στην ομάδα που συστήσαμε στη Ρώμη, όλοι μας επιδιώκουμε ένα σημαντικό στόχο που είναι η σταθεροποίηση της ε, Λιβύης ε, και στον Νίγηρα και στην Αλγερία και στην Τινησία θέλουμε σταθεροποίηση γιατί πιστεύουμε ότι για πολλές, πολλά χρόνια είχαμε εγκαταλείψει τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και σήμερα η ποιότητα ζωής ε, των ανθρώπων ε, στην Αφρική κυρίως στη Βόρεια Αφρική είναι τελείως ε, διαφορετική έχει βελτιωθεί κατά πολύ και εξ αυτού προκύπτει υποχρέωση της Ιταλικής κυβέρνησης έχουμε υποχρέωση έτσι ώστε και χώρες ε, όπως και το Τσάντ και η Τινησία να συνεργαστούν με μας ε, και με διεθνείς ε, οργανισμούς. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να μας βοηθήσετε. Ειλικρινά δεν θέλω να είμαι επιθετικός, αλλά εγώ ως ε, Ιταλός πολίτης, όχι ως νομάρχης, ως Ιταλός πολίτης συμμετέχω και η δική μου χώρα συνεισφέρει στα Ηνωμένα Έθνη για να ακούμε έναν ε, διευθυντή των Ηνωμένων Εθνών που αντί να ασχοληθεί με αυτά που του ζητάμε εδώ και πολύ καιρό, αυτά που ζητάμε από τους ε, διεθνείς υπαλλήλους να πάνε στη Λιβύη και να πάνε αλλού, τι κάνει, καταγγέλουν. Καταγγέλουν και δεν ξέρω κατά πόσον ε, το βράδυ κοιμούνται ήσυχοι για την αλληλεγγύη σε εισαγωγικά την οποία έχουν επιδείξει. Ο πρόεδρος Μωράης, ευχαριστώ πολύ κύριε Μορκόνε. Αντιλαμβάνεστε ότι αντιμετωπίζουμε πίεση χρόνου. Αν θα ήθελαν οι κύριοι ε, Φιλόρη και Πικέ να συμβάλλουν ώστε να μπορέσουμε να, απαντήσουμε, να απαντήσετε με λίγες φράσεις ο καθένας. Σας παρακαλώ, ναι. Πόσο χρόνο μου δίνετε κύριε Πρόεδρε? Ε, λίγα λεπτά. Είχα αντιληφθεί ότι αυτό θα συμβεί, αλλά έχουμε και ακρόαση. Πρώτα ε, ο κύριος Φιλόρη, να με συγχωρείτε, αλλά δεν μπόρεσα να κατανοήσω ορισμένες παρεμβάσεις ε, λόγω του ότι η μετάφραση δεν προλάβαινε να σας παρακολουθήσει. Euh, simplement une mise au point, s'il vous plaît, et je l'ai déjà, nous l'avons. Έχουμε κάτι πανάληψη πει και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους κόλπους της ε, συνέλευσής σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί κέντρα κράτησης στη Λιβύη. Κέντρα κράτησης, συμφωνούμε όλοι, πρέπει να κλείσουν. θα για να το επιτύχουμε αυτό. Να γνωρίζετε ότι η συνεργασία με οργανισμούς όπως IOM κλπ. Κάνουμε προσπάθειες για να επιτύχουμε το κλείσιμο των κέντρων αυτών και την αντικατάστασή τους από ένα σύστημα ανοιχτών κέντρων και να είναι σαφές λοιπόν αυτό. Δεν χρηματοδοτούμε κέντρα κράτησης στη Λιβύη. Δίνουμε χρήματα στους εταίρους μας, στον IOM και στον HCR, για να βελτιώσουν όσο μπορούν την μοίρα των ε, μεταναστών που κρατούνται στα κέντρα αυτά αναλαμβάνοντας δράσεις για την φροντίδα υγείας για την βελτίωση των συνθήκων υγιεινής, για παράδειγμα, και ιδίω για να συμβάλλουμε ώστε να μπορούν να εγκαταλείψουν τα κέντρα αυτά οι μετανάστες και πρόσφυγες από την αρχή του χρόνου μπορέσαμε να βγάλουμε έτσι χίλια πρόσωπα από τα κέντρα κράτησης χίλιες μικρές νίκες τις οποίες οφείλουμε να χαιρετήσουμε και αυτό έγινε με την πλήρη υποστήριξή μας το πρόβλημα είναι ότι για την ώρα οι λιβικές αρχές που διαχειρίζονται τα κέντρα αυτά δεν δέχονται να κινηθούν. Ο Υπατσαρμοστής για τους πρόσφυγες και ο IOM ζητούν να αντικασταθούν με ανοιχτά κέντρα. Και πιστεύω ότι το έχει κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την αποστολή που έχει στείλει στη Λιβύη θα έχει σίγουρα ταχθεί υπέρ αυτού. Στο μεταξύ πρέπει να βρούμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους επιτόπου και αυτό κάνουμε. Συμφωνούμε επίσης σχετικά με το ότι η λιβική ακτοφυλακή δεν έρεται στο ύψος των αναγκών, των περιστάσεων. Δεν δείχνει τον αναγκαίο επαγγελματισμό. Και για αυτό το λόγο επίσης σκοπεύουμε να τους εκπαιδεύσουμε. Και σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αυτής έγκυται στην διασφάλιση ανθρώπινης μεταχείρισης των μεταναστών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ισχύοντος διεθνούς δικαίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρο, συγγνώμη που σας πιέζω ε, χρονικά ε, και σας παρακαλώ να περιοριστείτε σε ορισμένα ε, βασικά. Εσείς, κύριε Πίκετ, αν είναι δυνατόν, ε, περιοριστείτε κι εσείς σε λίγα βασικά. Ναι, θα είμαι σύντομος, είχα το ίδιο πρόβλημα προφανώς με ε, το σύστημα, αλλά ε, για να είμαι σαφής, λαμβάνουμε υπόψη πολλά από τα όσα είπατε, συμφωνούμε με τις ανησυχίες που εκφράσατε απέναντί μας για τα κέντρα κράτησης, όπως είπε ο κύριος Φιλωρή, η ίδια η τη εκπρόσωπος στις 12 Σεπτεμβρίου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι θέλει να κλείσουν τα κέντρα κράτησης και κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρακινήσει τις ε, λιβικές αρχές να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Χρειάζεται να συμβάλλουμε να δημιουργηθούν εναλλακτικές επιλογές για την κράτηση των μεταναστών. Αυτά, σε αυτά συμβάλλουμε μέσω της χρηματοδότησης ανοιχτών κέντρων, όπως περιέγραψε ο κ. Φιλωρή, και την ενίσχυση των οικειοθελών επιστροφών. Το ξαναλέω δεν θα δεχόμαστε οποιαδήποτε άλλη βασική αρχή εκτός από αυτήν, ούτε άλλωστε οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Δεν πρόκειται για επαναπρόθεση, πρόκειται για οικειοθελείς επιστροφές. Ποια είναι η προτεραιότητά μας, ήταν μια από τις ερωτήσεις που μας κάνετε. Η προτεραιότητα της ΥΠΑ είναι η διάσωση ανθρώπινων ζώων και να προστατεύσει τους ανθρώπους και να δημιουργηθούν νόμιμες οδοί για την μετακίνησή τους προς την Ευρώπη όσων μεταναστών βρίσκονται στη Λιβύη και χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεύτερο βέβαια, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα παράτυπης μετανάστευσης. Εντός της Λιβύης υπάρχουν 700-800 άνθρωποι σε αυτήν την κατάσταση. Πρόκειται δηλαδή για μια ανθρωπιστική κρίση εν δυνάμει που ενδέχεται να επιδεινωθεί. Πρόκειται μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με κάθε μηχανισμό που διαθέτουμε. Και αυτά σας περιγράψαμε με τους συναδέλφους μου εδώ. Συνεργαζόμαστε με τις λιβικές αρχές, με την αναγνωρισμένη διεθνώς κυβέρνηση, η οποία είναι ασθενής κυβέρνηση. Με έλλειψη δηλαδή, έλλειψη ικανότητα ελέγχου όλη τη επικρότητα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στη χώρα αυτή. Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση αυτή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τα όσα συμβαίνουν στη Λιβύη. Α είμαστε πολύ ξεκαθαροί από αυτού. Και μέσα στο πλαίσιο τη συνεργασία μα αυτή, έχουμε άλλωστε και μια διαρκή συζήτηση όπου επισημαίνουμε στις αρχές αυτές τα προβλήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων σαν αυτά που συζητήσαμε και εδώ μαζί σας σήμερα. Τελευταίο σχόλιο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταθεροποιήσει την Λιβύη. Η θέση της ΥΠΑ εκπροσώπου είναι 100% υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας που στηρίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Βρίσκεται σε αδιέξοδο για την ώρα ή βρισκόταν σε αδιέξοδο μέχρι ότου ανέλαβε ο νέος εκπρόσωπος τον οποίον υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο πολιτικά αλλά και επιχειρησιακά με τεχνογνωσία, για παράδειγμα σε θέματα εκλογών, σε θέματα δημιουργίας θεσμών, σε εκπαίδευση για την δημιουργία θεσμών, διαμεσολάβηση μεταξύ των, των διαφόρων φορέων στην Λιβύη. Είναι βέβαια βαρύ έργο αυτό, αλλά κάτι στο οποίο δεσμεύεται απολύτως, είπατε εκπρόσωπος. Μάλιστα τούτη την εβδομάδα έχει πολλές συναντήσεις με Λίβιους εκπροσώπους για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Πριν αποχωρήσουν οι προσκεκλημένοι μας, τους οποίους ευχαριστώ βεβαίως, θα ήθελα να πω για τα μέλη. Βεβαίως ήταν συναισθηματικά φορτισμένη η συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη μας για τα όσα είπαν και να μην υπάρξει παρανόηση. Υπάρχει ανησυχία που εκφράζεται από τα μέλη και εγώ θα το επιβεβαιώσει αυτό κύριε Βερζιά, συναντήσαμε μέλη της Λιβικής Αυτοφυλακής και με τους Ιταλούς όλοι επενδύουμε πολύ προσπάθεια στα όσα συμβαίνουν στην Λιβύη και έχουμε εντονότητα τις ανησυχίες. Δεν πρόκειται για μια εφάπαξ συζήτηση. Τα θέματα αυτά τα συζητούμε ολόκληρη την ημέρα σήμερα. Έγινε και η Αφρικανική διάσκεψη υπό την αιγίδα του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου. Κάνουμε σημαντικότατη προσπάθεια. Και γι' αυτό εκφράζεται και τόσο μεγάλη ανησυχία και υπάρχει τέτοια συναισθηματική φόρτιση. Επιθυμώ να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών για την προσπάθεια που κάνουν και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Μορκόνε. Θέλετε κάτι να πείτε εσείς κύριε περισιά. Α, βλέπω ότι είναι διαδικαστικό αυτό που ζητείτε. Πρόεδρε, μια που με αναφέρατε πολλές φορές στα σχόλιά σας, θα συμφωνήσω όλα με μια διαφορά. Η Λιβική Ακτοφυλακή δεν ελέγχει παρά ένα μικρό μόνο μέρος της Λιβικής ακτής. Αυτό μας υπόθηκε και μας το επανέλαβαν. Το ζήτημα είναι ποιος ελέγχει την Λιβική επικράτεια και σε αυτό δεν έχουμε απάντηση. Γιατί ακούμε ένα σωρό πράγματα που οδηγούν την κοινή γνώμη να πιστέψει ότι πολύ ωραία συνεργαζόμαστε με τη Λιβική κυβέρνηση, άρα γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στη Λιβύη. Ε, δεν ισχύει αυτό. Ναι. Ε, ναι. πράγματι γνωρίζουμε πώ αναλύεται η κατάσταση στην Λιβύη. Αντιληφθήκαμε και τι συμβαίνει και με τα κέντρα κράτηση κλπ. Στην... Ε, Μπορεί να συνεχίσει κανεί, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε φτάσει στο τέλο τη προσπάθεια και θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τι και του συναδέλφου για την συνδρομή του σήμερα και να ευχαριστήσω και του προσκεκλημένου μα. θα συνεχίσουμε την συζήτηση. Βεβαίως ευχαριστώ και την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και την Προεδρία που μας παρεχώρησε έξτρα χρόνο. Σας ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε στην ακρόασή μας. Thank you Λοιπόν, για την ε, ακρόαση θα αρχίσουμε αμέσω. Όσοι παραμένετε λοιπόν για αυτή την ακρόαση, ωραία. Οι υπόλοιποι παρακαλώ να φύγετε ησύχω. Είναι ακρόαση με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φίλων. ΦΑΜ. Παρακαλώ την Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών να έρθει εδώ μαζί μου.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 Uh, um, Συναδελφοί, αν είμαστε όλοι έτοιμοι, μπορούμε να αρχίσουμε και ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε. Θέλω να αρχίσω εισάγοντας κάπως το θέμα εδώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω εδώ την πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών μαζί μας. Όπως ξέρετε συνάδελφοι, η ακρόαση αυτή έχει να κάνει με κάτι που ετοιμάζουμε, ένα σχέδιο έκθεσης τώρα, γιατί το λέω ακρόαση, ε, επειδή έχουμε εδώ και την Επιτροπή Γυναικών. Πρόκειται λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Θα θυμόσαστε ότι το 2010 ξεκίνησε αυτή η ιστορία και άρχισε να ισχύει τον Ιανουάριο η οδηγία. Οι χώρες μέλη έπρεπε να υποστηρίξουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 είναι μια ευκαιρία για τους ηγητές της ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής Γυναικών να δούνε πώς έχει κατάσταση σήμερα όσον αφορά την αμοιβαία εναγνώριση που σημαίνει ότι όταν υπάρχει μια εντολή προστασία σε μια χώρα αυτή πρέπει να αναγνωρίζεται και από την άλλη. Θα ακούσουμε λοιπόν τους οι που θα μας παρουσιάσουν τα κύρια ζητήματα. Και πρόκειται για την κυρία Πώς και την κυρία Χιμένες Μπεθερίλ. Συνεπώς, θα δώσω το λόγο στις εισηγήτριες. Τι λέτε. Α, ή να σας δώσω εσά τον πρόεδρο. Α, μου λέτε εγώ να συνεχίσω. Καλά. Εντάξει, θα συνεχίσω εγώ τότε. Οπότε, θα δώσω το λόγο πρώτα στη Σοραγιά Πόστ. Για πέντε λεπτά παρακαλώ. Και μετά στη Τερέσα για άλλα πέντε λεπτά. Παρακαλώ λοιπόν, πέντε λεπτά για την παρουσίασή σου. Ευχαριστώ πολύ Κλοντ. Ναι, είχα την τιμή να δουλέψω στην έκθεση αυτή όσον αφορά την υλοποίηση της οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία, η οποία εφόσον λειτουργήσει θα ε, σώσει Ζωέ ανθρώπων που είναι θύματα βία, ανδεκογενειακή βία ή άλλη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία λοιπόν που όπω σας είπα σώζει χιλιάδε ζωέ. Διαπιστώσαμε όμως με την συνεισηγήτριά μου, την Τερέσα Χιμένες Μπεθερίλ, ότι μόνο 7 τέτοια ευρωπαϊκά εντάλματα προστασίας έχουν εκδοθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα. Κάτι το οποίο δείχνει ότι μέχρι τώρα ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οι χώρες μέλη έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους αρκετά στα σοβαρά. Οι αξιωματούχοι που έρχονται σε επαφή με τα θύματα δεν γνωρίζουν τίποτα πολύ συχνά για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Οι διαφορές οργανώσεις ούτε και αυτές. Τα θύματα ούτε και αυτά. Άντε και μόλις μεταβίας αναγνωρίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εθνική τους προστασία και αλλού στο εξωτερικό αν θέλουν να ταξιδέψουν και να πάνε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Συνεπώς εμείς στο σχέδιο έκθεσής μας διατυπώνουμε διάφορα αιτήματα σε πολλές σελίδες και λέμε τι βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε, μεταξύ των οποίων είναι και τα εξή. Κάνουμε έκκληση στι χώρε μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατάλογο αρχών που είναι υπεύθυνε κάθε φορά για την έκδοση και την αναγνώριση τη Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία. Και θέλουμε και ένα κατάλογο κεντρικών αρχών που στέλνουν ή παραλαμβάνουν τέτοιες ευρωπαϊκές εντολές προστασίας και να είναι εύκολο να έχει πρόσβαση σε τέτοια εντολή κάθε άτομο που νιώθει ότι απειλείται. Και θεωρεί ότι έχει ανάγκη από την Ευρωπαϊκή αυτή εντολή προστασίας. Να γίνεται εκτίμηση για το κάθε άτομο με, την, με βοήθεια και με μέτρα στήριξης εφόσον ε, κάποιο ζητήσει Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Επίσης, οδηγεί στις χώρες μέλη για να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν άτομα με οι ειδικέ ε, ανάγκες που ζητούν εντολή τέτοια προστασίας. Κάνουμε έκκληση επίσης στην Επιτροπή και στις χώρες μέλη να θέσουν ένα χρονοδιάγραμμα στις αρμόδιες αρχές τους προκειμένου να εκδίδουν ευρωπαϊκές εντολές προστασίας και να μην παρατείνουν αβεβαιότητα και να δώσουν οδηγίες στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να ενημερώνουν επαρκώς τα θύματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετά από την οποία θα υπάρξει απόφαση για εντολή προστασίας. Επίσης, ζητούμε περισσότερη συνεργασία με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, προσέγγιση βάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάρτιση όλων των αξιωματούχων που εμπλέκονται με τα θύματα και αυτό σε τακτική βάση. Και να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί ορθά να ακολουθήσει μια ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, αστυνομία, ποιος. Επίσης κάνουμε έκκληση στις χώρες μέλη να ε, προχωρήσουν σε εκστρατείες συνειδητοποίησης και εκστρατείες γενικότερα κατά της ενδοικογενειακής βίας ή γενικότερα βία σε βάρος των γυναικών με συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και μια που ήμουν εισηγήτρια εκ μέρους της ΛΥΜΠΕ είχα και τις δικές μου ανησυχίες όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας των προσώπων. Με την πρόσφατη άφηξη προσφύγων και τούντων ε, άσυλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται περισσότερο με την εξωτερική πτυχή. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ενδοικογενειακή βία και την αντιμετωπίζουμε λίγο πολύ όλοι. Φτάνει να κοιτάξει κανείς τα στοιχεία για να ξέρει ότι χρειάζεται προστασία ε, των ε, ατόμων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην γίνονται θύματα διαπροσωπικής βίας. Μια στις τρεις γυναίκες ήταν θύμα ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας. Μία στις πέντε ε, έχει γίνει θύμα παρενόχλησης. Μία έξι γυναίκες ήταν θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Το μέγεθος φαίνεται και από την εξαρτία που κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, όπου οι γυναίκες πια έρχονται και μοιράζονται τις εμπειρίες τους για την ε, απειλή αυτή που υπέστησαν και την ε, βία από πλευράς ε, αντρών της, σεξουαλική δηλαδή παρενόχληση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ανασφάλεια στις γυναίκες εξαιτίας τέτοιων φαινομένων. Ευχαριστούμε η Τερέσα Χιμένε Μπεθερίλη έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω στην άλλη συγκίτρια την κυρία Σοράγια Πόστ, για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Πολύ καρποφόρα. Συνεργαστήκαμε προκειμένου να βελτιώσουμε την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας και προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα μέσο το οποίο αποτελεσματικά θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των θυμάτων ε, εγκληματικών πράξεων. Και λέει όλα, γιατί συνήθως την εντολή αυτή προστασίας τη βλέπουμε σαν κάτι που μπορεί να προστατεύσει τις γυναίκες από την ενδοοικογενειακή βία. Και όντως, κυρίως γυναίκες ζητούν αυτήν την εντολή προστασίας, επειδή είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Αλλά υπάρχουν και άλλα θύματα, είτε τρομοκρατίας, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε ο οποίος απειλείται από κάποιον άλλον που μπορεί να ζητήσει αυτή την εντολή προστασίας. Φτιάχτηκε λοιπόν για άτομα τα οποία είναι θύματα εγκλημάτων και μπορούν να ζητήσουν εντολή προστασία σε μια χώρα και αυτή να ισχύει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ήμουν λοιπόν εισηγήτρια στην Επιτροπή Γυναικών όταν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ισπανική Προεδρία ζητήθηκε η προσπάθεια αυτή. Η υποδοχή ήταν πολύ θερμή και οι προσδοκίες ε, βέβαια ακολούθησαν. Γι' αυτό και όντως πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να έχουμε ένα νέο μέσο, πιο δυναμικό μηχανισμό που να απομακρύνεται από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που είχαμε στην αρχή. Κάτι το οποίο αποτρέπει συχνά τα θύματα να προσφύγουν σε τέτοιους μηχανισμούς όπως είναι η εντολή προστασία. Σκεφτείτε κάποιος ο οποίος πηγαίνει σε μια χώρα που δεν γνωρίζει τη γλώσσα, πώς θα αποδείξει ότι όντως χρειάζεται προστασία. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό αυτόματα από τη μία χώρα στην επόμενη χώρα να υπάρχει, να εμφανίζεται αυτή η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, οπότε να μην χρειάζεται το θύμα να κάνει απολύτως τίποτα. Έχει εκδοθεί στη χώρα του μία τέτοια ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, όταν βρεθεί σε άλλη χώρα, η άλλη χώρα αυτόματα το βλέπει ότι χαίρεται της προστασίας αυτής. Πολύ βασικό για το χώρο μας ε, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Χρειάζεται ένας μηχανισμός δικαστικής συνεργασίας λοιπόν. Το μέσο αυτό που είχαμε μέχρι τώρα στη διάθεσή μας δεν είχε αποτελέσματα. Και τώρα είπαμε ότι μόνο 10 γυναίκες είχαν καταφέρει να πετύχουν τέτοια προστασία εξαιτίας αδικογενειακής βίας. 7 μόνο. 4 στην Ισπανία, 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο και μία εντολή προστασίας έχουν εκδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα. Εντάξει, δεν ζήτησαν αυτήν την προστασία πολλές γυναίκες, ναι, αλλά μόνο 7. Μόνο 7. Δεν ε, θέλω να πω περισσότερα, αλλά κοιτάξτε, πριν από λίγο στη χώρα μου, πριν από μια εβδομάδα, μια Γερμανίδα πήγε στο Καστεγιόν, που είναι κοντά στη Βαλένθια, και δολοφόνησε μια άλλη η Γερμανίδα. Ε, δεν έγινε καταγγελία. Πρόκειται λοιπόν για άτομα ε, τα οποία μπλέχτηκαν σε αυτό το έγκλημα και είναι από διαφορετική χώρα. Και το έγκλημα έγινε σε διαφορετική χώρα. Άρα χρειάζεται ο μηχανισμός αυτός. Το 2011 λοιπόν άρχισε να ισχύει η οδηγία αυτή, αλλά δυστυχώς από τότε δεν συγκεντρώθηκαν αρκετά στοιχεία για να δούμε πώς χρησιμοποιείται αυτός ο μηχανισμός. Δεν έχουμε σημεία αναφοράς δηλαδή. Οπότε το σχέδιο το δικό μας βασίζεται σε μία μελέτη της ε, δικιάς μας υπηρεσίας κοινοβουλευτικών ερευνών. Δεν υπάρχει κεντρικό μητρό για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Πώς να την αξιολογήσουμε λοιπόν. Είναι περίπλοκη επίσης η εφαρμογή της οδηγίας από τις εθνικές αρχές και άρα είναι πολύ δύσκολο το θύμα να καταλάβει. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο επίσης για τα πιο ευάλωτα άτομα. Τέλος υπάρχει παραπληροφόρηση για τις εθνικές αρχές. Δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση. Δεν εφαρμόζεται η εντολή προστασία σε όλες τις χώρες, οπότε και η Κομισιόν που να ξέρει τι γίνεται. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στο συντονισμό και στην επικοινωνία μεταξύ χωρών μελών για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Το θύμα δεν έχει στη διάθεσή του μετάφραση. Για ένα τέτοιο διασυνοριακό εργαλείο καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Το θύμα θα πρέπει να έχετε δυνατότητα να ενημερώνετε κατάλληλα στη γλώσσα του και να μπορεί έτσι να ζητάει η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Διαπιστώσαμε όμως ότι υπάρχουν ε, πολλά κενά και γενικά δεν υπάρχει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς ε, τα θύματα στις διάφορες χώρες. Και είναι πολύ κακό να μην υπάρχει ενημέρωση για την προστασία των θυμάτων. Κάθε φορά που μετακινείται από μία χώρα σε άλλη ένα θύμα κινδυνεύει να βρεθεί σε ένα ξένο νομικό σύστημα, σε γλώσσα την οποία να μην γνωρίζει, άρα καθίσταται ακόμα πιο ευάλωτο το θύμα από ό,τι ήταν ήδη. Και δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη δυνατότητα και σίγουρα όχι για άτομα με ειδικέ ανάγκες. Για να υπάρξει λοιπόν αποτελεσματική προστασία θα πρέπει η διαδικασία για την έκδοση και την ε, υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας να γίνεται γρήγορα και να βρούμε τρόπο ώστε άμεσα να εκδίδονται τέτοιες εντολές προστασίας, να ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες. Άλλο σημαντικό πράγμα είναι ο συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των κεντρικών αρχών για την προστασία των θυμάτων και την αποτελεσματικότητα της εντολής αυτής. Ζητούμε λοιπόν από τις χώρες μα να δημιουργήσουν ένα σύστημα εθνικού μητρώου για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας και να γίνεται και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει ένα σύστημα ευρωπαϊκού μητρώου όπου θα συγκεντρώνονται όλες τι πληροφορίες από όλες τις χώρες μέλη για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Οι δικαστικές νομικέ αδυναμίες στην σημερινή οδηγία αντιμετωπίζεται εφόσον τα διάφορα μέσα προστασίας του θύματος που διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδυαστούν. Για παράδειγμα, η οδηγία για την οποία ήμουν εισηγήτρια εγώ και τώρα εφαρμόζεται, που είναι η Γενική Οδηγία για το δικαίωμα στην προστασία και την προστασία των θυμάτων από εγκληματικές πράξεις. Τέλος, η κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να δίνει πληροφορίες, ε, να φροντίζει για κατάρτιση των αρμοδίων αρχών και των επαγγελματιών, ε, νομικών και άλλων. Με τη βελτίωση αυτή πιστεύω ότι τα θύματα θα έχουν πιο εύκολα πρόσβαση στην εντολή προστασίας και θα την χρησιμοποιούν όταν τους έχουν εξηγήσει καλά περί τίνος πρόκειται, πώς εκδίδεται, πώς εφαρμόζεται κτλ. Και έτσι τα θύματα κάθε εγκληματική πράξης θα μπορούν να προστατεύονται και να αποφεύγουν να γίνουν θύματα δεύτερη φορά εξαιτία τη ελληπούς πληροφόρηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χιμένες Τεσσερίν. Θα δώσω το λόγο στα μέλη των επιτροπών. Όσοι εξημών επιθυμείτε να λάβετε το λόγο, αλλά όχι πάνω από δύο λεπτά ο καθένας. Και πρώτα οι σκιώδεις συγητές. Ρωτώ εάν θέλετε να μιλήσετε. Πρώτη, πρώτη κύριε Τσέτμαρ. Έχετε το λόγο. Ναι. Και μετά θα ακολουθήσουν άλλα μέλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το κείμενο της εκθέσεως έχει καλώς Και οι δύο συνεισηγήτριες τα πήγαν πολύ καλά και τις ευχαριστώ. Στην έκθεση νομίζω περιλαμβάνονται και όλα τα σχόλια που είχα κάνει εγώ ίδιος στην πρώτη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, διότι η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία είναι ένα σημαντικό μηχανισμό και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλήρω σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να εξασφαλιστεί ότι από πλευρά χωρών μελών και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαφημιστεί εντό εισαγωγικών αρκετά, δηλαδή θύματα βίων πράξεων να έχουν εύκολη πρόσβαση στον μηχανισμό αυτό. Χαίρομαι λοιπόν για το σχέδιο που έχουν υποβάλει οι δύο συναδελφοί μου. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε μου, θα καταβάλω προσπάθεια να αναπτύξω κάποια θέματα με περισσότερη λεπτομέρεια. Αλλά πάντως το κείμενο στο σύνολό του με ικανοποιεί. Σα ευχαριστώ και πάλι. Η κυρία Βλανκεβιτσιούτε. Κύριε Ορτασούν, Ευχαριστώ. Πρώτα επιθυμώ να ευχαριστήσω τις συνεισηγήτριες για τη θαυμάσια δουλειά που έκαναν. Βρισκόμαστε προς τα πράγματι σε ένα σημαντικό μηχανισμό. Το είπαν και οι δύο εισηγήτριες. Από τότε όμως που καθιδρύθηκε το 2015 μόνο 7 φορές έχει χρησιμοποιηθεί, 7 δηλαδή εντολές προστασίας έχουν εκδοθεί. Ωστόσο η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να υπάρχει σε μεγάλους αριθμούς, άρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Να έρθω σε ορισμένα από τα θέματα που νομίζω ότι θα πρέπει να διορθωθούν στο, ε, στο μηχανισμό. Πρώτα θα ήθελα να πω, άλλωστε ορισμένα από αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση. Απογοητευόμαστε λίγο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή. Τα ίδια όταν μιλούσαμε και για την οδηγία κατά του, του, της λαθροδιακίνησης. Δεν είχαμε έκθεση εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ αυτή είναι υποχρεωμένη να διαθέτουν σχετικές πληροφορίες, να ξεκινούν τις διαδικασίες για παραβίαση κατά των χωρών μελών, εφόσον δεν εφαρμόζονται σωστά οι μηχανισμοί αυτοί και μέχρι τώρα δεν έχουν καν συλλέξει τα δεδομένα. Από τότε που ε, ισχύει ο μηχανισμό αυτό. Άρα πρέπει να του λάβουν σοβαρά υπόψη του. Δηλαδή, εννοώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο, έχουμε ζήτημα εναρμόνιση επιπέδων προστασία σε ορισμένε χώρε μέλη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρει η έκθεσή μα. Ορισμένε χώρε μέλη δεν περιλαμβάνουν ποινική δίωξη κατά του λεγόμενου stalking, δηλαδή τη επίμονη παρενόχληση. Και βεβαίω ε, υπάρχουν τέτοια θύματα. Ε, άλλο ένα θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Άλλο πρόβλημα του ΕΠΟ, δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία, είναι η έλλειψη ενημέρωση για τα θύματα. Θα χρειαστεί λοιπόν να γίνουν κάποιε εκστρατείε ευαισθητοποίηση για να εξηγηθούν τα του μηχανισμού. Θέλουμε να στηρίξουμε επίση την ιδέα τη παροχή εκπαίδευση σε αξιωματούχου αστυνομία, δημοσίων αρχών, καθώ και ασκούμενου νομομαθεί ή αυτούς ε, που ασκούν το επάγγελμα του μαχόμενου δικηγόρου ή του δίκαστου. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πρόκειται για σημαντικό μηχανισμό, δεν έχει όμως επαρκή προώθηση από τις χώρες μέλη. Για να επιτευχθεί αυτό, ευχαρίστω θα συνεργαστούμε με τις δύο συνεισηγήτριες για να φτιάξουμε μια στέρεη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Merci ε, ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε. Λίγα λόγια για να τονίσω και εγώ τον θαυμάσιο χαρακτήρα της εκθέσεως των δυο συναδέλφων που είναι πλήρης, παρουσιάζει ε, τις ε, δυσκολίες, τους λόγους ε, αποτυχίες και αδυναμίες και την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμού για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων. Για αυτό το μηχανισμό προστασίας ήδη ήμουν εισηγήτρια εγώ από το 2010. Είχαμε κάνει αγώνα τότε για να φτιαχτεί ένας μηχανισμός που θα είναι στέρεος, λογικά δομημένος, που θα επιτρέπει εν τέλει πέρα από το ίδιο το αντικείμενο, δηλαδή την εντολή προστασίας ε, των θυμάτων, δηλαδή που κυρίως είναι γυναίκες, να ενσαρκώσει αυτό που σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να υπάρξει μια συνέχεια δικαστική προστασίας των προσώπων που μετακινούνται σε άλλη χώρα μέλος. Ήταν η πραγματική πεμπτουσία της ιδέας της Ευρώπης και θυμούμε ότι τότε είχα χαιρετήσει και μάλιστα με ενθουσιασμό τον μηχανισμό συνεργασίας, την πρόοδο σε ό,τι αφορά την πρόληψη, σε ό,τι αφορά την βοήθεια προς τα θύματα, όταν είχαμε υιοθετήσει τότε τον σχετικό μηχανισμό. Εγώ πάντως εκπλήσωμαι και θλίβομαι που βλέπω ότι μόνο 7 εντολές προστασίας έχουν εκδοθεί. Ούτε πιστεύω στα μάτια μου που βλέπω τον αριθμό αυτό. Ασφαλώς η ποικιλία, οι διαφορές των εθνικών ε, δικαιικών τάξεων οδηγούν πιθανότατα στον περιορισμό αυτό αριθμό, η ελληπή συνεργασία μεταξύ χωρών μελών. Διερωτώ με, υπάρχει παρουσία του Συμβουλίου σήμερα η απάντηση δεν θα ευρεθεί εδώ, διότι εδώ όλοι συμφωνούμε. Όλες συμφωνούμε, όλες κατανοούμε την έννοια, τη σημασία του ε, κειμένου και τι πρέπει να μπορεί να κάνει η Ευρώπη για τους πολίτες και, τις, ε, των δύο φίλων. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι προκλήσεις. Προτείνουμε λύσεις και δύο μόλις μέρες πριν από την ε, Διεθνή ημέρα αγώνα κατά της βίας κατά των γυναικών Όλοι μιλούν για την απολύτως αναξιοπρεπή κατάσταση ε, που σημειώνεται σε ορισμένες χώρες μέλη. Πρέπει να, κάνουμε, να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια διαφήμισης όπως είπαν άλλοι. Αλλά πρέπει να υπάρξει και μια συγκεκριμενοποίηση στο επίπεδο των χωρών μελών. Ασφαλώ και υπάρχει προσθέμενη αξία του μηχανισμού αν όμως κανένα δεν το χρησιμοποιεί, τότε ποιον εξυπηρετεί. Και τέλος τι εξυπηρετούμε εμείς εδώ. Εμείς, οι θεσμοί. Εάν συζητούμε επί μήνες για την δημιουργία ενός μηχανισμού που τελικώ δεν εξυπηρετεί κανένα. Θα λάβουμε απάντηση, διότι άλλωστε οι αρμόδιοι να δώσουν απαντήσεις δεν είναι καν εδώ σήμερα η απάντηση δεν πρέπει να αναζητηθεί εδώ, διότι εδώ όλες είμαστε πεπισμένες για την αξία του μηχανισμού της εντολής προστασίας. Αλλά πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η προστασία των θυμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ρε, κυρία Μπουλάν, κύριε Θα δώσω λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Είμαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη. Ε, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή τη θαυμάσια έκθεση, ε, πολύ συνοπτική και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Όλα αυτά που συμπεριλαμβάνει η έκθεση. Επίσης, και εμείς ε, ανησυχούμε για το ότι ε, δεν εφαρμόζεται ικανοποιητικά αυτό το τόσο σημαντικό εργαλείο. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σωστή εφαρμογή και των δύο εργαλείων και της οδηγίας και του κανονισμού. Η σωστή λοιπόν εφαρμογή είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Για μας αυτά αποτελούν προτεραιότητα. Όσον αφορά στην οδηγία. Τους τελευταίους μήνες ε, ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το να υπάρξει σωστή μεταφορά αυτού του εργαλείου και πρέπει να σας πω ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει αυτή την οδηγία στην νομοθεσία τους πλήρης λοιπόν μεταφορά σε εθνική νομοθεσία από όλα τα κράτη-μέλη και με αυτήν την ενημέρωση από πλευρά ε, κρατών μελών νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στην έκθεση και στην εφαρμογή αυτού του εργαλείου κυρίως για το πώς τα θύματα και άλλα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο μπορούν να κάνουν χρήση της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας. Το 2018 θα καταθέσουμε σχετική έκθεση. Επίσης, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας όλες τις ανησυχίες που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και στην ε, ε, διάδοση πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Γι' αυτό λοιπόν ως Επιτροπή αποφασίσαμε να έχουμε μια διαδικτυακή πύλη ε, με που αποκαλείται η γωνία των θυμάτων, Victims Corner, Εκεί θα αναφέρονται οι εθνικές αρμόδιες αρχές ε, αλλά και όλες οι άλλες πληροφορίες ε, που αφορούν στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας που θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι και εύκολα προσπελάσιμη για όσους θέλουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Ε, ευρωπαϊκή εντολή προστασία σε ε, θέματα αστικού δικαίου, αλλά τώρα θέλουμε ε, να υπάρχει ευρωπαϊκή εντολή προστασία και για ποινικά θέματα οποτεδήποτε συναντιόμαστε με εθνικούς εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με θα συζητάμε το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα στις 21 Ιανουαρίου έχουμε προγραμματίσει μία ε, συνάντηση ψηλοεπιπέδου με εθνικού εμπειρογνώμονες για θέματα θυμάτων και εκεί θα συζητηθεί ακριβώς αυτό το θέμα. Δηλαδή θα ε, ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της συζήτησης ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συζητήσω με τα κράτη-μέλη για το πώς ε, τα θύματα και άλλοι που βρίσκονται σε κίνδυνο μπορούν πραγματικά να αποφεληθούν από αυτό το τόσο σημαντικό εργαλείο. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Και τώρα έχουν το λόγο οι δύο συνεισηγήτριες. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω. Πράγματι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει μόνο τέσσερις, ε, με συγχωρείτε, επτά, επτά τέτοιες ε, εντολές. Αλλά ε, εντωμεταξύ έχουν κατατεθεί περίπου 40.000 σε εθνικό επίπεδο, αλλά μόνο σε ευρωπαϊκό. Άρα δηλαδή Αυτά καταδεικνύουν ότι πράγματι κάτι πρέπει να γίνει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Επιτροπή ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες ήταν πρόθυμη να προσφέρει επιπρόσθετες πληροφορίες. Ε, συνεργαστήκαμε και νομίζω το θέμα αυτό ε, πρέπει πραγματικά να αναχθεί σε πρώτη προτεραιότητα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εκτεθειμένοι στη βία. Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές και την Τερέζα γιατί δουλέψαμε εξαιρετικά χωρίς ε, κανένα απολύτως πρόβλημα. Η κυρία Χιμένες. Ευχαριστώ και εγώ. Και ευχαριστώ πολύ τη Σωράγια Πόστ. Τα πόλα όλα στην αρχή. Το μόνο που θέλω να κάνω τώρα είναι να ευχαριστήσω τους σκιώδες εισηγητές και να εκφράσω την ικανοποίησή μου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκει σιγά σιγά στοιχεία γιατί δεν είχε υλικό στη διάθεσή της και αυτό είναι ένα άνοιγμα για τα θύματα προκειμένου να μπορέσει να ισχύσει η οδηγία. Η κυρία Κρίκ έχει δίκιο όταν ε, λέει πως δημιουργήθηκαν πολλές προσδοκίες και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι δεν πήγε καλά. Μα έλειψε η πολιτική βούληση. Αυτό δεν πήγε καλά. Γι' αυτό και δεν λειτουργήσε όλη η αλυσίδα. Ούτε η πληροφόρηση υπήρξε, ούτε κατάλληλη κατάρτιση στην αστυνομία κλπ. κλπ. Νομίζω ότι το θύμα έχει το πρόβλημα ε, και το θύμα φοβάται, σιωπά και γι' αυτό δεν μιλάει. Εμείς μπορεί να πούμε, ναι, αλλά το θύμα δεν κινείται. Δεν υπήρξαν περισσότερες εντολές προστασίας γιατί το θύμα φοβάται να ταξιδέψει, κάθεται στη γωνίτσα του. Ναι, αλλά ίσως ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε, να πάμε και να του πούμε ότι μπορεί να ταξιδέψει, ότι αν έχει φίλους, οικογένεια, λούσα, άλλη χώρα, μπορεί να το κάνει μπορεί να έχει την προστασία αυτή και αλλού. Τι θα κάνω αν πάω σε άλλη χώρα, σκέφτεται το θύμα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να στηρίζουμε περισσότερο το θύμα και να προσπαθήσουμε να το βοηθήσουμε και να το ενημερώσουμε γιατί πρέπει να έχει κάποιο κίνητρο για να προχωρήσει και να ζητήσει έκδοση ε, εντολής προστασίας. Στη χώρα μου τέσσερις μόνο. Και όμως είμαστε πρωταθλητές στη Γαλλία, καμία μία στην Ιταλία, στη Γερμανία. Μας εκπλήσουν αυτά τα αποτελέσματα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ Τέρεσα. Και τις δύο σκιώδεις εισηγητρίες. Η προθεσμία είναι η 7η Σεπτεμβρίου για την υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέρφους και της ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής Γυναικών για την παρουσία τους εδώ σήμερα. Οπότε τελειώσαμε με αυτήν την κοινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ και την Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών και τα μέλη της. Τώρα, συνεχίζει η Λίμπε. Και πάμε στο σημείο 12. Εδώ έχουμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, μια σύντομη μελέτη. Περιμένω να έρθουν εδώ οι συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο 12 στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευση, σχετική μελέτη που θα μας παρουσιαστεί σήμερα για την παράνομη εργασία μεταναστών από τρίτε χώρες. Έχουμε εδώ τον κύριο Τζούλιαν Τάγκερμαν, ο οποίος είναι ερευνητής συνεργάτης και πολιτικός αναλυτής στο Γερμανικό Εθνικό Σημείο Επαφής ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. Θα ενημερωθούμε από την μελέτη αυτή ποιες είναι οι τάσεις, θα γίνει κάποια σύγκριση και θα δούμε με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει κυρώσεις κατά των εργοδοτών, για παράδειγμα. Και επίσης θα εξετάσουμε και νόμιμες ε, οδούς έλευσης μεταναστών τρίτων χωρών. Θα συζητήσουμε για το τι δεν εφαρμόζεται ικανοποιητικά και τι γίνεται με τις περιπτώσεις μεταναστών οι οποίοι παράνομα ζουν στις χώρες μας. Κύριε Τάγκερμαν, έχετε το λόγο 10-15 λεπτά και μετά θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις με τους ευρωβουλευτές. Μισή ώρα συνολικά. Ναι. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθετε και έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκλησή σας και για την προσφώνηση. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθερών που δίνει στο European Migration Network την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα της μελέτης μας για την παράνομη απασχόληση ε, υπηκών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγομαι Τάγκερμαν και είμαι ερευνητής στο ε, τμήμα ερευνών του Γερμανικού Γραφείου για πρόσφυγες και είμαι και contact point επομένω για σχετικά θέματα. Υπενθυμίζω ότι, ότι η ΕΜΕΝ έχει 28 σημεία επαφής είτε σε δημόσιες αρχές, είτε σε πανεπιστήμια, είτε σε ε, αντιπροσωπείες διαφόρων διεθνών οργανισμών. Η μελέτη που θα σας παρουσιάσουμε βασίζεται στις συμβολές 23 εθνικών ε, σημείων επαφής το 2016 σύμφωνα με ένα ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε έκθεση η οποία βρίσκεται στον σύνδεσμο που βλέπετε, καθώς και οι εθνικές συμβολές. Χάρη στην, λόγω της ε, ε, Συνεργασία αυτή δεν θα μπορέσω να πω σε λεπτομέρειε. Θα προσπαθήσω ωστόσο να σα δώσω μια συνολική επισκόπηση για την κατάσταση στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. Γιατί ο ή εμένα αποφάσισε να ασχοληθεί με την παράνομη απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών. Αφενός διότι ω γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει εντολή να αντιμετωπίσει την ε, παράνομη ε, απασχόληση και ιδίω μέσω τη οδηγία του 2009 παρόλο που, λοιπόν, που υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για την παράνομη απασχόληση που οδηγεί σε μείωση των εισφορών, μείωση των ε, φόρων, ε, ανταγωνισμό από την πλευρά των των τρίτων χωρών και ούτω καθεξής και βεβαίω θίγονται και τα κοινωνικά δικαιώματα των προσώπων αυτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται ανάλυση των μέσων και μέτρων που βρίσκονται στο επίπεδο των χωρών μελών για τον εντοπισμό των προβληματικών περιοχών και να διευκολυνθούν μέσω βέλτιστων πρακτικών. Η μελέτη θεωρεί την παράνομη απασχόληση υπηκών τρίτων χωρών ως απασχόληση η οποία δεν ε, σέβεται το υφιστάμενο δίκαιο. Έχουμε εξετάσει λοιπόν την παράνομη απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν πλέον τις προϋποθέσεις για να, παραμένουν, να διαμένουν μόνιμα στις ε, χώρες μέλη. Από την άλλη μεριά εξετάζει η μελέτη επίσης την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν νόμιμο καθεστώς αλλά απασχολούνται παρανόμως, δηλαδή εκτός του πλαισίου του δικαίου για την εργασία οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες τρίτη ε, ε των χωρών δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. Λαμβάνονται υπόψη ορισμένα σημαντικά μέτρα, μέτρα πρόληψης ε, τη παράνομη απασχόλησης υπηκότητα ε, των χωρών, εντοπισμό ιδίω μέσω επιθεωρήσεων, κυρώσει για εργοδότες που απασχολούν παράνομα υπηκότητα των χωρών και τέλος τις επιπτώσεις για τους ίδιους τους επικόστον των τρίτων χωρών. Έχω ορισμένα ε, συγκεκριμένα περιστατικά ή ορισμένες συγκεκριμένες ενδείξεις για, τις, ε, για τα αποτελέσματα της ε, μελέτης μας. Όσο ό,τι αφορά τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες μέλη για να μειώσουν την παράνομη απασχόληση πριν αυτή αρχίσει. Υπάρχουν πρώτα κάποια κοινά μέτρα αυτά που στρέφονται κατά των εργοδοτών ή πιθανών εργοδοτών και αυτά που στρέφονται ενδεχομένω κατά των επικών τρίτων χωρών. Οι περισσότερε χώρε μέλη που συμμετέσχουν στην ε, έρευνα είπαν ότι κάνουν ε, προσπάθειες εκστρατείε συνειδητοποίησης. Οι περισσότερες χώρες μέλη δίνουν πληροφορίε και κυρίως μέσω ιστοσελίδων και στι δύο ομάδε ενδιαφερομένων. άλλε χώρες μέλη διαθέτουν νομοθεσία που υποχρεώνει του εργοδότε να ενημερώνουν τι αρμόδιες αρχέ για την έναρξη και για την περαίωση τη ε, σχέση εργασία με τον ε, υπηκό τρίτων χωρών και υπάρχουν και συγκεκριμένες νομοθεσίες ορισμένε χώρε μέλη για του υπηκό τρίτων χωρών. Ορισμένε χώρε μέλη τονίζουν επίση ότι συμφωνίε εταιρική σχέση με οργανώσει είτε συνδικάτα, οργανώσει δηλαδή εργοδοτών είτε συνδικάτα, λαμβάνουν υπόψη την προσπάθεια αντιμετώπιση τη παράνομη απασχόληση. Τι απαντήσει του οι χώρε μέλη εντοπίζουν και διάφορου παράγοντε επιτυχία από την πλευρά των εργοδοτών. Βλέπουμε, για παράδειγμα, πρώτα το αποτέλεσμα αποτροπής που μπορούν να έχουν οι κυρώσει, εφόσον θα μιλήσουμε αργότερα για τι κυρώσει κατά των εργοδοτών. Δεύτερον, την καθίδρυση συνεργασιών είτε επισήμων είτε ανεπισήμων μεταξύ διαφόρων φορέων και οργανώσεων στο εθνικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, τονίζεται ότι η ενδυνάμωση των εργαζομένων που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα με πληροφορίες και με νομικές υπηρεσίες μπορεί να είναι ένας θετικός παράγοντας για να αποφευθεί η εκμετάλλευση των προσώπων αυτών από τους ασυνείδητους εργοδότες. Και αυτά γίνονται συχνά από συνδικάτα ή μη κρατικέ οργανώσεις εάν δεν λειτουργήσει τελικώ η πρόληψη και υπάρξει παράνομη απασχόληση υπηκό τρίτη της χώρας, ε, εκεί αρχή περιβλέκεται το πράγμα. Τώρα, εκεί διαπίστωσαν χώρες μέλη ότι, ή μάλλον η έρευνα, ότι είναι διαφορετική η ε, αντιμετώπιση. Αφενός υπάρχουν επιθεωρήσεις εργασίας που κάνουν επιτόπου επιθεωρήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως αυτά οι επιθεωρήσει αυτές ανατίθεται και σε άλλες αρχές, όπως για παράδειγμα στι τελωνιακές αρχές, στην περίπτωση της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Αυτό όμως συνολικά για την παράνομη εργασία. Η Φιλανδία ως μόνη χώρα μέλος έχει ειδική μονάδα που ασχολείται με την εργασία αλλοδαπών. Οι επιθεωρήσει γίνονται κυρίω στη βάση αναλύσεων κινδύνου που εντοπίζουν τους πλέον επικίνδυνους τομείς και αυτό προβλέπεται στο άρθρο 14 της σχετικής οδηγίας και εκτελείται σε όλες τις χώρες μέλη, μέλη εκτός από μία. Οι περισσότερες χώρες μέλη προβλέπουν επιθεωρήσεις σύμφωνα με εθνικά κριτήρια, για παράδειγμα λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης ή το μερίδιο δαπων απασχολούμενων στην συγκεκριμένη επιχείρηση, ο καθεξής ξεκινά συχνά από καταγγελίες του κοινού οι περισσότερες χώρες μέλη έχουν και ειδική hotline, ειδική τηλεφωνική γραμμή δηλαδή για καταγγελίες. Σε άλλες χώρες μέλη οι επιθεωρήσεις πηγαίνουν επί τόπου, συζητούν με απασχολούμενους και διαπιστώνουν τα γεγονότα καθώς και τη σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Σε ορισμένες χώρες μέλη εξετάζονται και τα έγγραφα των ε, απασχολουμένων. Σε ορισμένες χώρες μέλη μας είπαν ότι ο αριθμός του προσωπικού που κάνει τι επιθεωρήσει αυτέ είναι πάρα πολύ περιορισμένο και επομένω οδηγεί στην έλλειψη αποκάλυψη τέτοιων περιπτώσεων. Επιθυμεί κανεί βέβαια να γνωρίζει το μέγεθο του προβλήματο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε ανεπαρκή δεδομένα και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι οι στατιστικέ δεν είναι πλήρω διαθέσιμε και ότι οι χώρες μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες για την συλλογή των δεδομένων αυτών. Επομένως δεν είναι εγγυημένη η συγκρισιμότητα. Πέραν αυτού, και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να το έχει κανείς υπόψη, λόγω του ότι υπάρχει και μια κρυφή φύση του φαινομένου αυτού, δεν υπάρχουν πλήρη διαφανή στοιχεία της απασχόλησης των υπηκών τρίτων χωρών, παρά μόνο σε περιπτώσεις επιβολής του νόμου που και αυτές επηρεάζονται από μεγάλο αριθμό παραγόντων. Τα δεδομένα που έχουμε λοιπόν είναι πάρα πολύ επιλεκτικά. Μπορούμε λοιπόν να συναγάγουμε μόνο κάποια προκαταρκτικά συμπεράσματα και ένα από αυτά είναι ότι η κατανομή των μη εντοπισμένων περιπτώσεων σε όλες τις χώρες μέλη είναι πολύ άνηση μεταξύ των χωρών μελών. Βλέπουμε επίσης ότι οι παράνομα απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι κυρίως άνδρες μεταξύ 25 και 35 ετών εργάζονται σε μικρές ή μεσές επιχειρήσεις σε τομείς που απαιτούν χαμηλου επιπεδου προσόντα, τουρισμός, εστιατόρια, οικοδομή. Μεταξύ των περιπτώσεων, εφόσον εντοπιστούν τέτοιες και ε, κρυθεί υπεύθυνο εργοδότης, υπάρχει η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Είναι πολύ διαφορετικέ κυρώσεις που επιβάλλονται ένα χώρα μέλο. Βλέπετε την ε, διαφάνεια, τον αριθμό των χωρών μελών που επιβάλλουν ε, κυρώσεις για την παράνομη απασχόληση παράνομων βγικών ε, τρίτων χωρών και ούτω καθεξής. Βλέπετε επίσης εδώ ότι συνήθως οι χώρες μέλη επιβάλλουν πρόστιμα. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα πρόστιμα και το επίπεδο των προστήμων είναι ποικίλει πολύ μεταξύ χωρών μελών και εξαρτάται από το καθεστώς του απασχολουμένου και από την βαρύτητα της παράβασης. Άλλα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες μέλη είναι και ποινές φυλάκισης και κατάσχεση των κερδών, κλείσιμο της επιχείρησης, προσωρινό ή οριστικό, και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Ρωτήσαμε επίσης πόσες χώρες μέλη κάνουν υπολογισμό της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα αποτέλεσματα. Ισχυρό, ισχυρή είναι η αποτροπή των προστήμων και χρηματικών ειναι πολυ διαφορετικα τα αποτελεσματα η ισχυρη ειναι η αποτροπη των προστημων και χρηματικων κυρωσεων Άλλες χώρες θεωρούν ότι οι σχετικές τιμές είναι πολύ, ποινές, συγγνώμη, είναι πολύ ήπιες και επομένως η αποτρεπτικότητα είναι χαμηλή. Ένα βασικό το οποίο προκύπτει από τις ε, συνεισφορές των χωρών μελών είναι ότι ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των κυρώσεων δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την αυστηρότητα της νομοθεσίας, αλλά περισσότερο από την εφαρμογή επιβολή δηλαδή των κυρώσεων. Οι χώρες μέλη τονίζουν επίσης ότι υπάρχουν προκλήσεις. Τέσσερις χώρες μέλη εντοπίζουν το monitoring, την αποκάλυψη και την απόδειξη των παράνομων απασχολήσεων. Και σχετικό με αυτό είναι και η συνεισφορά μιας χώρας μέλου, μέλους ότι είναι ανεπαρκείς οι πηγές ή μάλλον είναι ανεπαρκείς οι πόροι που επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατάστασης. Έχουν εντοπιστεί βεβαίως στην έρευνά μας και καλές πρακτικές όπου υπάρχει εξορθολογισμένη ε, προσπάθεια στο, εθνικό επίπεδο, αλλά βεβαίως και αποτελεσματικός μηχανισμός υποβολής καταγγελιών, από πλευρά δηλαδή των απασχολουμένων, που επιτρέπει τότε την επιβολή κυρώσεων κατά των εργοδοτών. Τέλος, μια σύντομη ματιά στο τι συμβαίνει στους υπηκόους των τρίτων χωρών όταν διαπιστώνεται ότι αυτοί απασχολούνται παρανόμως. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων κράτηση, επιβολή προστήμων, ε, να θεωρηθούν, να ταυτοποιηθούν δηλαδή ως θύματα λαθροδιακίνησης, να χάσουν το δικαίωμα παραμονής ή τέλος μπορεί να χάσουν όπως είπα το, το δικαίωμα της διαμονής. Η μελέτη περιλαμβάνει και πολλές case studies και υπορισμένους συσχετισμούς ε, περιστάσεων και ανάλογα με τη χώρα μέλος όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο πρόσωπο η έκβαση μπορεί να είναι διαφορετική. Ωστόσο η μελέτη, ή μάλλον οι case studies, οι μελέτες περιπτώσεων δηλαδή δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις σύμφωνα με την ομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους ο υπήκος τρίτης χώρας μπορεί να αντιμετωπίσει απόφαση επιστροφής 23 χώρες μέλη το λιγότερο πιθανό είναι να λάβει εν τέλει καθεστώς παραμονής και απασχόλησης. Να τακτοποιηθεί δηλαδή η περίπτωσή του. Αυτό συμβαίνει σε εννέα μόνο χώρες μέλη από αυτές που συμμετέσχουν στην έρευνα. Η έκβαση για τους επικοστήτων τρίτων χωρών είναι και η δυνατότητα να ζητήσουν αποζημίωση για μη καταβληθέντα, για δεδουλευμένα. Μπορούν δηλαδή να στραφούν κατά του εργοδότη εφόσον έχουν σύμβαση εργασίας, ισχυρά σύμβαση εργασίας. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα να υποβληθούν καταγγελίες κατά των εργοδοτών. Ορισμένες χώρες μέλη μας λένε ωστόσο ότι σπάνια συμβαίνει αυτό στην πράξη και αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Η διστακτικότητα των επικών τρίτων χωρών να συνεργαστούν με τις ε, δημόσιες αρχές διότι φοβούνται ότι θα απελαθούν και λόγω του κρυφού χαρακτήρα της απασχόλησης αυτής συχνά αποτυχαίνει αυτό. Επίσης προβλήματα γλωσσικών φραγμών. Ιδίω το ζήτημα της λήψης πληροφοριών είναι σημαντικό για να μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να προβούν στις αναγκαίες ε, δράσεις. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν και μάλλον 12 χώρε μέλη ε, θεωρούν ότι πρέπει να γίνει συστηματική πληροφόρηση των υπηκών τρίτων χωρών για τα δικαιώματα που απορρέουν από την οδηγία. Σημαντικό επίση για του υπηκού τρίτων χωρών για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν του μηχανισμού καταγγελιών και να καταγγέλουν του εργοδότε του. Η πληροφόρηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη με χαμηλά κατόφλια και υπάρχουν καλές πρακτικές όπως δείχνει η μελέτη επίσης παροχή συμβουλών από μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή από εργατικά συνδικάτα. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, η μελέτη εντοπίζει τα εξής ε, πορίσματα είχε γίνει μια μελέτη το 2015 και επιβεβαιώθηκαν τα συμπεράσματα, δηλαδή ότι θα πρέπει ε, να υπάρξουν περισσότερες δράσεις κατά των, ε, της παράνομης απασχόλησης υπηκών τρίτων κρατών. Εγώ θα αναφέρω δεικτικά κάποια από αυτά τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Πρώτον, ε, πρόσβαση στους μηχανισμούς καταγγελίας και στην ενημέρωση για τα δικαιώματα. Δεύτερον, βελτίωση του αριθμού των περιπτώσεων όπου εντοπίζεται παράνομη απασχόληση. Αυτό σε πολλά κρατημέλη έχει σχέση με το προσωπικό ε, και αυτά βεβαίως ε, συμβαδίζουν και με τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Ε, αποφασίσαμε και ότι η επιβολή των κυρώσεων είναι πολύ σημαντική για να είναι αποτρεπτική, αποτρεπτικός παράγων. Αυτό είναι ένα καθοριστικό βήμα για να περιοριστεί η παράνομη απασχόληση υπηκών τρίτων χωρών. Εξάλλου πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι ότι δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Την ώρα που ολοκληρώθηκε η μελέτη, το 2016, 18 κράτη-μέλη είχαν ήδη υιοθετήσει ή επρόκειτο να υιοθετήσουν νέα νομοθεσία επί του θέματος. Και με αυτά θα ήθελα να ολοκληρώσω. Ε, ελπίζω να μπορέσω να δώσω έτσι κάποια γενική εικόνα σε αυτές τις 125 σελίδες ε, της μελέτης και βεβαίως ε, με μεγάλη χαρά να απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ για την ε, ομιλία σας. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις εθνικότητες ε, αυτών των ε, ε, παράνομα απασχολούμενων ε, ε, μεταναστών των τρίτων, υπηκών τρίτων χωρών. Από πού έρχονται και ποιοι είναι οι τομείς, οι χαρακτηριστικοί τομείς, κλάδοι μάλλον με συγχωρείτε, όπου απασχολούνται οι υπήκοοι τρίτων κρατών. Παραδείγματος χάρη στη δική μου τη χώρα τα εστιατόρια ε, με εθνικά χαρακτηριστικά είναι εκείνα όπου απασχολούνται περισσότερο οι η αυτοί. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, δύο ομάδες ανθρώπων. Αυτοί που έρχονται ως ε, πρόσφυγες και δεν τους χορηγούν το άσυλο και αυτοί παραμένουν και υπάρχει μια άλλη ομάδα που προέρχονται, έρχονται από άλλες χώρες που δεν ζήτησαν ε, άδεια παραμονής γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα την πάρουν έτσι κι αλλιώ. Υπάρχουν λοιπόν δύο ομάδες υπηκών τρίτων κρατών και δεν ξέρω, εσείς κάνετε τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Παραδείγματος χάρη στη δική μου τη χώρα, τη Σουηδία, ε, πάρα πολλοί ε, που δεν έχουν χαρτιά είναι εκείνοι που απορρίφθηκε η αίτησή τους ασύλου, δεν ε, επιστρέφουν στην πατρίδα τους, ε, παραμένουν σε εμά, ακόμα και αν τους πληρώνουν οι δικές μας οι αρμόδιες αρχές. Προτιμούν να παραμείνουν στη χώρα μας. Και στη Σουηδία, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να είναι κανείς παράνομος, κυρίως το χειμώνα. Και μετά έχουμε και αρκετούς που έρχονται από χώρες όπου είναι αδύνατον να αποκτήσει κανείς άσυλο. Αυτοί έρχονται, παραμένουν στη χώρα και κανείς δεν ξέρει πόσοι τελικά είναι. Ε, διερωτώ με, έχετε εσείς ε, κάποια εικόνα ε, σχετικά με αυτές τις ομάδες ανθρώπων, οι μεν έχουν χαρτιά, οι άλλοι ίσως όχι. Και τι είδους προστασία μπορεί να υπάρχει για άτομα που δεν έχουν χαρτιά όσον αφορά στα δικαιώματά τους όχι μόνο σχετικά με την οδηγία περικυρώσεων, αλλά και με άλλα δικαιώματα που αφορούν στους εργαζόμενους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. κυρία Τσινίτση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δόκτωρα Τάγκερμαν για την ομιλία του. Εγώ είμαι Ιταλίδα οι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, ανάμεσα αυτές δεν είναι η Ιταλία. Όμως εμείς έχουμε κάνει σημαντική δουλειά για να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε την εκμετάλλευση ε, εργαζομένων από τρίτες χώρες, κυρίως στον γεωργικό τομέα και στον τομέα της διατροφής. Υπάρχει λοιπόν η εκμετάλλευση αυτών των ε, εργαζομένων ε, και αυτή η εκμετάλλευση γίνεται κυρίως από εγκληματικές οργανώσεις. Και θέλω να ρωτήσω, εντοπίσατε να υπάρχει κάτι παρεμφερές και σε άλλες χώρες, δηλαδή εγκληματικές οργανώσεις που να χειρίζονται, που να είναι ε, υπεύθυνε για αυτό το φαινόμενο. Κάτι άλλο, σε σχέση με την προστασία και την πρόληψη. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχουν προληπτικά μέτρα που να αφορούν και στην εργασία και στους εργαζόμενους. Σας κάνω αυτή την ερώτηση γιατί εδώ πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία σιγά σιγά αναδύεται, δηλαδή ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης. Παραδείγματος χάρη στον γεωργικό τομέα και τον τομέα των ε, τροφίμων ε, όπου διαπιστώνουμε αυτό το φαινόμενο θεωρώ ότι ο καταναλωτής ε, θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και αν θέλετε και να έχει εκπαιδευτεί σωστά. Όχι μόνο για το θέμα της υγείας ε, σε σχέση με την παραγωγή του προϊόντος, αν είναι οικολογικό ή όχι, αλλά θα πρέπει ο καταναλωτής να είναι ενημερωμένος και για την ηθική διάσταση της παραγωγής ε, και κάτι άλλο που αφορά στις ε, καταγγελίες. Είπατε και ισχύει ότι η αποκάλυψη περιπτώσεων εκμετάλλευσης είναι πολύ δύσκολη γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για να γίνουν οι έλεγχοι. Ε, μήπως υπάρχουν όμως ε, και άλλοι λόγοι. Άλλοι λόγοι είναι παραδείγματο χάρη ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν αποκαλύπτουν ε, τέτοιου είδου φαινόμενα γιατί φοβούνται ότι ενδεχομένως μετά να βρεθούν σε κέντρα κράτησης ή να χάσουν το δικαίωμα διαμονής στη χώρα. Υπάρχουν λοιπόν πρωτοβουλίες που να βοηθούν ε, τους εργαζόμενους για να ε, προβαίνουν σε καταγγελία και μετά να ακολουθούν όλες οι άλλες φάσεις ε, που ακολουθούν μετά από την, ε, από την καταγγελία. Η κυρία Τζιν Λάμπερτς. Ευχαριστώ και εγώ. Συγγνώμη που έχασα την αρχή και ίσως κάποια από αυτά που ρωτήσω να έχουν ήδη υποθεί και απαντηθεί. Θέλω να έρθω σε κάποια θέματα που έθιξαν και συνάδελφοι για ξεχωριστούς τομείς. Γιατί από όσο θυμάμαι εγώ την νομοθεσία αυτή, αυτό που έκανε ήταν ότι επικε... ζητούσε μάλλον από τις χώρες μέλη να επικεντρωθούν στην ε, επιθεώρηση εργασίας. Ρωτάω λοιπόν, αυτός ο στόχος ισχύει ή οι χώρες μέλη επειδή ασχολήθηκαν ε, με διάφορα ζητήματα κάποια τα άφησαν απ' έξω. Ήταν δηλαδή η στρατηγική αποτελεσματική. Ξέρω ότι κάποιες χώρες και δικιά μου ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα με τις άδειε για τους εργοδότες και τα λοιπά, αλλά δεν το κάνουν. Και όσον αφορά τους πόρους που δίνονται, όταν τα κοιτάξαμε, γιατί εγώ συμμετέχω και στην Επιτροπή Απασχόλησης, όταν ρωτάτε τις χώρες να σας πούν για την επιθεώρηση εργασίας, τελικά δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, ότι τους πόρους δεν τους βάζουν στην επιθεώρηση εργασίας. Τώρα το θέμα της ανάκτησης των μισθών κλπ. Κατά πόσο τα παίρνουν τα χρήματα αυτά οι εργαζόμενοι. Αρχικά είχαμε πει ότι οι χώρες μέλη έπρεπε να πληρώσουν αυτά τα οποία έπρεπε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και μετά να τα ανακτήσουν από τους εργοδότες. Δεν μπήκε στην οδηγία τελικά. Υπάρχουν όμως χώρες που πληρώνουν τα χρωστούμενα και μετά ανακτούν τις οφειλές από τους ίδιους τους εργοδότες ή τελικά αφήνουν τον κόσμο να παλεύει, να πάρει αυτά τα οποία δικαιούται τα δουλεμένα του. Και κάτι άλλο που ρώτησα και συνάδελφοι για τα στοιχεία που διατηρούν τα κράτη-μέλη για αυτά. ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Υπάρχουν στοιχεία και για τον αριθμό των ανθρώπων που απασχολούνται με αυτόν τον τρόπο. Ρωτήθηκε κάτι για την ε, κατανομή αναφύλλο ή αναεθνικότητα. Υπάρχουν καθόλου τέτοια στοιχεία. Τέλος. Υπάρχουν χώρες μέλη όπου τρίτα μέρη. Αν δηλαδή οι ίδιοι εργοζόμενοι δεν θέλουν να πάνε να καταγγείλουν μια περίπτωση που γίνεται εκμετάλλευση, μπορεί ένα τρίτο μέρος να προσφύγει στη δικαιοσύνη ανταυτών. Ευχαριστώ. Κύριε Λεμπρετό. Ο κύριος Λεμπρετό, συγγνώμη. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ρμάν για τα όσα μας είπε. Το θέμα που συζητάμε είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για ξένους εργαζόμενους παράνομους που έρχονται από άλλες χώρες ε, από ό,τι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε μας αλλάζει συνήθως τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με τους αποσπασμένους. Αλλά πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα λέμε ότι πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις στους εργοδότες που εκμεταλλεύονται την ε, ταλαιπωρία και την κακομεριά του κάθε εργαζόμενου και μας λέτε ότι γίνονται βελτιώσεις σε πολλές χώρες μέλη. Ωραία, καλό είναι αυτό. Όμως, πιστεύω ότι πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις και στους ίδιους τους παράνομους εργαζόμενους, τους ξένους, εφόσον δέχονται παράνομα μια θέση απασχόλησης. Και αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, γιατί έχουμε πολλή ανεργία στις χώρες μας. Οπότε είναι αναγκαίο να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο της παράνομης εργασίας με όλες τις, τις μορφές. Δυστυχώς, ομολογείται ότι παρά τις καλές προθέσεις δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την παράνομη εργασία των ξένων, γιατί σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν αρκετοί επιθεωρητές εργασίας, π.χ. Οπότε, Κατόπιν τούτου, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, αυτή τουλάχιστον είναι η δικιά μου, ότι στις χώρες μέλη τι γίνεται. Πρώτον, είναι προφανές ότι η Συμφωνία Σέγγεν που άνοιξε πλήρως τα σύνορα βοήθησε την έλευση των μετανοστών και έφερε σε δύσκολη θέση πολλές χώρες. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάπτυξε μια πολιτική λιτότητας που ανάγκασε πολλές χώρες να μειώσουν το περιθώριο ελεγμών που είχαν ε, τις δημόσιες δαπάνες τους ας πούμε, με αποτέλεσμα σε πολλές χώρες η ε, επιθόρηση εργασίας έχει αποδεκατεστεί. Και τρίτον, πολύ εύκολο είναι να κλαίμε πάνω στις συνέπειες, αλλά τις αποφάσεις εμείς τις πήραμε για αυτές. Και τρίτον, μια ερώτηση. Μήπως υπάρχουν ε, λόμπι πίσω από όλους αυτούς τους ελιγμούς για να υποφεληθούν από την παράνομη εργασία. Γιατί για πολλούς εργοδότες οι παράνομοι αυτοί οι εργάτες κοστίζουν πολύ λιγότερα από ότι οι καταγεγραμμένοι νόμιμοι κτλ. Εσείς τι λέτε για το ρόλο των λόμπις και των πολυεθνικών. Μήπως τελικά επηρέασαν πολύ τα πράγματα και έτσι φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κύριε Τάγερμαν, για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας. Μία-μία θα τις απαντήσω. Πρώτον, για τις εθνικότητες και τους τομείς. Πράγματι, έχουμε κάποια δεδομένα για κάποιες χώρες μέλη. Δεν έχουν στοιχεία όμως όλες οι χώρες συνολικά. Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε να κάνουμε την ανάλυση. Βασιζόμαστε στις χώρες που έδωσαν στοιχεία. Όσον αφορά τους τομείς, ισχύει αυτό που είπα στην παρουσίασή μου, στις χώρες μέλη για τομείς που απαιτούν χαμηλές δεξιοτεχνίες ισχύει για τομείς όπως είναι ο οικοδομικός, η ε, τροφοδοσία κλπ. Δεύτερη ερώτηση. Ρωτάτε για τις διαφορές ανάμεσα στους πρόσφυγες που δεν πήραν το καθεστώς αυτό και υπηκός τρίτων χωρών που μπαίνουν στις χώρες για να βρούνε μια δουλειά, όποια και αν είναι. Στη μελέτη δεν κάναμε τη διάκριση αυτή. Αυτό που μπορώ να σας πω από τη Γερμανία και με την κύριο που έχει αναλάβει το γερμανικό τμήμα της μελέτης, δεν είχαμε πολύ κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης για αυτό το θέμα και δεν έχουμε και εμπειρικές μελέτες για να μπορέσουμε να διακρίνουμε αυτές τις δύο κατηγορίες και να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους. Άρα λοιπόν υπάρχει έλλειψη γνώσης εδώ. Για το θέμα των δικλείδων ασφαλείας. Το ρωτήσατε πολλές φορές. Φυσικά η οδηγία για τις κυρώσεις τους εργοδότης προβλέπει διαδικασίες προσφυγών που ξεκινάει η χώρα μέλος. Και στη μελέτη είδαμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί προσφυγής εφαρμόζονται με διαφορετικούς τρόπους στις χώρες μέλη. Υπάρχει η καλή πρακτική στο Βέλγιο, για παράδειγμα, που στην επιθεώρηση εργασίας υπάρχει δυνατότητα υπήκοη τρίτης χώρας με την εγγύηση ότι δεν θα τους ε, καταγγείλουν στη συνέχεια, ότι θα τους προστατεύσουν, ανώνυμα δηλαδή, να μπορούν να προσφύγουν κατά των εργοδοτών τους. Βρήκαμε ότι είναι πολύ πρακτικό αυτό. Διαπιστώσαμε όμως ότι γίνονται και πολλά από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και συνδικάτα που προσφέρουν βοήθεια με κέντρα όπως γίνεται στη Σουηδία και την Αυστρία για να μην ονομάσω παρά δύο μόνο χώρες μέλη όπου υπάρχουν κάποιοι χώροι συγκεκριμένοι και μπορούν οι εργαζόμενοι που δεν έχουν χαρτιά να πάνε και να ζητήσουν συμβουλές και στήριξη για να προσφύγουν στη συνέχεια κατά των εργοδοτών τους. Το θέμα τώρα των εγκληματικών οργανώσεων, κατά πόσο δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα η μελέτη, δεν μπήκε σε αυτό, δεν είχαμε τέτοια ερώτηση. Από τις ισπανικές επαφές μας και οργανώσεις, μας είπαν ότι όλο και περισσότερο ασχολούνται με το θέμα. Για το θέμα της πρόληψης, όσον αφορά γενικά τον κόσμο, δεν ξέρουμε για εκστρατείες που να έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά θα μπορούσε να είναι τομέας δράσης αυτός. Και μετέχατε και μια άλλη ερώτηση που επανέλαβαν οι συνάδελφοι για τις τρίτες πλευρές κατά πόσο είναι σε θέση, ένα τρίτο μέρος δηλαδή, κατά πόσο είναι σε θέση να υποβάλει προσφυγή αντί του εργαζόμενου, κατά πόσο μπορεί να δράσει δηλαδή εκ μέρου των υπηκών τρίτων χωρών. Αυτό προβλέπεται στην οδηγία για τις κυρώσεις απέναντι εργοδότες και σε κάποιες χώρες μέλη γίνεται. Την άλλη σας ερώτηση δεν μπόρεσα να την απαντήσω στην έκθεση ότι βρείτε. Τώρα, σχετικά με τους ε, στόχους, ε, κατά πόσο τους πετύχαμε, πράγματι ε, τους πετύχαμε. Είναι ένα επιτυχημένο μοντέλο και πρέπει να σας πω ότι δεν εξετάσαμε την αποτελεσματικότητα των ε, επιθεωρήσεων, τουλάχιστον ε, όχι κάτω από το πρίσμα του αριθμού των υπηκών τρίτων χωρών οι οποίοι απασχολούνται παράνομα. Άρα δηλαδή η απάντηση ε, σε αυτή την ερώτηση είναι ότι ξέρετε αυτό δεν το μέσα στις έρευνές μας και γι' αυτό δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Ως προς τους πόρους, ορισμένα κράτη-μέλη μας είπαν ότι πράγματι οι πόροι δεν επαρκούν αλλά αυτό ετέθη από ορισμένα κράτη-μέλη και εν πάση περιπτώσει αυτή την απάντηση δεν την έδωσαν συχνά και αρκετά κράτη-μέλη. Όσον αφορά τα δεδομένα, ε, τα οποία κρατάνε τα κράτη-μέλη και τα χωρίζουν ε, αναφύλο και άλλα ε, χαρακτηριστικά και άλλες κατηγορίες, πράγματι ορισμένα κράτη κρατάνε, τηρούν τέτοια δεδομένα ε, διαχωρισμένες σε κατηγορίες, αλλά πάλι δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό, για να βελτιώνονται οι αναφορές. Και να πω και κάτι επ' αυτού. Όσο καλύτερες γίνονται οι αναφορές, ε, τόσο καλύτερες μπορούν να γίνουν και επιθεωρήσεις. Ε, τόσο καλύτερα στοχευμένες είναι επιθεωρήσεις ε, και τελικά τόσο καλύτερα προκύπτουν και τα δεδομένα. Είναι ένα είδος φαύλου κύκλου που προκύπτει. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι για να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων ή μάλλον αν βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων αυτομάτως αυξάνεται γενικότερα και όλη μας προσπάθεια. Ε, οι τελευταίες ερωτήσεις που έχω γράψει αφορούν στην ε, αντιμετώπιση των ίδιων των υπηκών ε, τρίτων ε, κρατών. Όπως αναφέρω στα συμπεράσματά μας, η νομοθεσία των κρατών μελών προβλέπει αποτελέσματα τα οποία μπορούν πράγματι να ερμηνευθούν ως κυρώσεις. Όμως ε, είναι σημαντικό για τους υπηκόους τρίτων κρατών να μπορούν να δράσουν και αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο αν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Δεν έχουμε μπει στο ερώτημα πόσοι υπήκοοι τρίτων κρατών έχουν επαρκή πληροφόρηση και πόσοι δεν έχουν όταν ε, ξεκινάνε μια παράνομη απασχόληση. Νομίζω όμως ότι στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να έχουμε κατά ότι ε, κάποιος μπορεί να δράσει μόνο εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε πότε ακριβώς ε, δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες. Ε, θα έλεγε κανείς ότι τελικά ε, πολλές φορές πληροφορίζονται αρκετά καθυστερημένα, αλλά για ορισμένους υπηκόους τρίτων κρατών αυτό είναι το πρώτο σημείο επαφής με κρατικές αρχές. Η Σλοβακία και η Γαλλία, παραδείγματο το κάνουν αυτό. Όσον αφορά το θέμα των ε, ομάδων πίεσης, σχετικά με την παράνομη απασχόληση των υπηκών τριτών κρατών. Αυτό δεν μας απασχόλησε στην έρευνα. Ε, δεν έχουμε πληροφορίες από αυτού. Ε, ελπίζω να απάντησα ικανοποιητικά στις ερωτήσεις σας. Αν όχι μπορείτε κάλλιστα βεβαίως να μου το επισημάνετε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Ευχαριστούμε και για τους συναδέλφους που σας υπέβαλαν τις ερωτήσεις. Όλα αυτά που είπατε ε, είναι ιδιαίτερα επικοδομητικά. Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Και τώρα σας ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, έχουμε άλλο ένα θέμα πριν περάσουμε στην ε, ψηφοφορία που είναι και το τελευταίο θέμα σήμερα της μέσης διάταξης είναι το σημείο υπερθμών 13 το επόμενό μας θέμα είναι ενημέρωση από τον εισηγητή για την Eurodac, αλλά δεν βλέπω την κυρία Μακοβέη να είναι στην αίθουσα. Δεν έχει έρθει ενδεχομένω ακόμα. Okay, so we're waiting for... Oh, nobody's interested, it's fine. Sorry, how many minutes? Well, she's coming. Νομίζω σε περίπου δύο λεπτά θα έρθει η κυρία Μακοβέη. Αυτό λοιπόν τον άπλετο χρόνο να τον χρησιμοποιήσετε για να κάνετε κάτι, αν θέλετε μπορείτε να διασκεδάσετε. Εγώ θα κοιμηθώ λιγάκι, είμαι πτώμα. You know. She said Uh, λοιπόν, σε δύο λεπτά θα είναι εδώ η κυρία Μακοβέη και θα μας ενημερώσει για τον τριμερή διάλογο σχετικά με τη Eurodac. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να περιμένουμε και μετά θα περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Ξέρω ότι ε, υπάρχουν ε, συνάδελφοι που έχουν έρθει εδώ ειδικά για την ψηφοφορία. Διακόπτουμε για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.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 Well, AUTHORWAVE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 au Conseil et la Commission. Non, non, je ne crois Where are we? 17. So, colleagues, um, we're going to. Ας αρχίσουμε, μάλλον ας επαναλάβουμε τώρα, ήρθε η για το θέμα υπαριθμών 13 και Αντιλαμβάνομαι βεβαίω ότι πλησιάζει και το τέλος της ημέρας. Ε, η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 17 και 45 και ορισμένοι συνάδελφοι έχουν έρθει ειδικά γι' αυτό, Άρα μια σύντομη παρουσίαση από ε, πλευρά της ηχηρήτριας για το Eurodac. Πρόκειται για αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac με εισηγήτρια την κυρία Μακοβέη η οποία θα μας ενημερώσει για την ε, πορεία του τριμερούς διαλόγου και ως γνωρίζετε το θέμα είναι μέρος του πακέτου μεταρρύθμισης και έχουν, για τις και μέχρι τώρα έχουν γίνει τρεις συναντήσεις τριμερούς διαλόγου, έτσι δεν είναι, στην Εστονική Προεδρία στη διάρκεια της Εστονικής Προεδρίας και νομίζω προβλέπονται άλλοι δύο τριμερείς διάλογοι μέχρι τέλους της Εστονικής Προεδρίας. Θα παρακαλέσω την κυρία Μακοβέη βέβαια να κάνει μια σύντομη παρουσίαση, μια σύντομη ανάπτυξη του θέματος γιατί όπως είπα 17 ε, και 45 προβλέπεται η ψηφοφορία. Αν θα θέλατε κυρία Μακοβέη. Πόσα λεπτά μου δίνετε κύριε Πρόεδρε. Πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά. Ναι, ναι, έχει καλώ. Εντάξει, μου φτάνουν. Όπως είπατε, έχουν γίνει τρεις συναντήσεις τριμερούς διαλόγου. Αύριο προβλέπεται άλλο ένα τριμερής διάλογο, αλλά αναβλήθηκε δυστυχώ για την επόμενη εβδομάδα. Μπορέσαμε να συμφωνήσουμε προσωρινώ για ένα αριθμό σημαντικών θεμάτων, ε, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα των χωρών μελών να ζητούν συγκρίσεις με δεδομένα ε, Eurodac στην βάση αλφα, αλφαριθμητικών δεδομένων ή βιομετρικών δεδομένων με πιο αποτελεσματική χρήση του χρόνου διότι γνωρίζετε ότι προβλέπεται και στον ε, παρόντα κανονισμό πρόσβαση της Europol στο EuroTac, αλλά για επιχειρησιακούς λόγους η Europol δεν είχε πρόσβαση τελικώς. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα για την χρήση τη κράτηση για την ταυτοποίηση του υπηκόου τρίτη χώρα. Είναι θέμα βέβαια εθνική νομοθεσία. Στο προήμιο λέμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι μέτρο ίστατη καταφυγής, η κράτηση δηλαδή, αφού εξαντληθούν τα άλλα. Επίσης προβλέπονται ειδικά πράγματα για τους ανήλικους. Αρχικά ισχύει το βελτιστό, το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου. Έχουμε ακόμη να επεξεργαστούμε πως θα αναγκαστεί κάποιος εφόσον ε, αρνείται να χορηγήσει βιομετρικά δεδομένα του προσώπου του. Έχουμε συζητήσει επίσης και κοντεύουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για την διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων. Εμείς έχουμε ζητήσει πέντε χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δέκα χρόνια και για το Eurodac επί του παρόντος προβλέπονται δέκα χρόνια, αλλά θα καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό κάπου ανάμεσα στα δύο αυτά όρια. Και εδώ χρειάζεται συμφωνία όλων των πολιτικών, ε, μάλλον διαφαίνεται συνένεση των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Περιμένουμε τώρα το Συμβούλιο Υπουργών, η Προεδρία μάλλον, να καταθέσει καθαρή κοινή θέση του Συμβουλίου για ορισμένα από τα θέματα αυτά και ολοκληρώνοντας θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις βαίνουν καλώς και εκτιμώ πολύ την ε, βούληση συνεργασίας που δείχνει η Εστονική Προεδρία θα ήθελα να ολοκληρωθεί η συμφωνία μέσα στα πλαίσια της Εστονικής Προεδρίας, πριν από την λήξη της δηλαδή, ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και ελπίζω θα μπορέσουμε, γιατί έχουμε ακόμα δύο συναντήσεις τριμερούς διαλόγου για τον Δεκέμβριο. Νομίζω τα είπα αρκετά σύντομα, έτσι κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακοβέη. Ρωτώ αν επιθυμούν οι σκιώδεις συγητές ή κάποιος σκιώδης συγητής να λάβει το λόγο. Α, η κυρία, η κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Κλοντ. Δεν έχουμε βέβαια πολύ χρόνο όπως εξήγησες. Απευθυνόμενοι στην ε, κυρία Μακοβέη θέλω να πω ότι μας θύμισε ότι σε ορισμένα θέματα έγιναν πρόοδοι, ότι με συνεργασία της Εστονικής Προεδρίας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε διαπραγματευτεί με πολύ θετικό τρόπο, είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε ένα σημαντικό θέμα που ανέφερε προηγουμένως άλλωστε η συναδελφός μου κυρία Μακοβέη. Υπάρχει συνένεση σχετικά με το ότι η Ευρωπόλ στο μέλλον θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε σύγκριση δεδομένων όχι μέσω κάτω χωρών χωρίς παρέμβαση δηλαδή τρίτων, αλλά απευθείας. Θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη ακόμα συζήτηση, ωστόσο, και δεν είμαι βεβαία ότι θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε, να, να κλείσουμε δηλαδή την δέσμη μέχρι τέλου τη Εστονική Προεδρία, για παράδειγμα, για την μείωση του ελάχιστου ορίου ηλικία για την λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εκεί είπαμε ότι χρειαζόμαστε πολύ ισχυρέ safeguards ε, υπέρ των ανηλίκων και αυτό σημαίνει βέβαια ότι αντιτασσόμαστε και στην κράτηση ανηλίκων καθώς και στην αναγκαστική λήψη δακτυλικών αποτιμάτων παιδιών. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική θέση του Κοινοβουλίου και εκεί θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω στον τριμήρη διάλογο. Εκεί όπου κατά την αντίληψή μου δεν βρισκόμαστε ακόμη προεπικείμενη συμφωνίας είναι για την διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων. Εμείς ως Επιτροπή έχουμε πει πέντε χρόνια για τα πρόσωπα που ζητούν άσυλο. Αυτό ήταν και μια σημαντική απόφαση της παρούσας Επιτροπής Θεμελιώδων Δικαιωμάτων. Από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένουν στα δέκα χρόνια. Παραπέμποντας μεταξύ άλλων και στους κανόνες της Συμφωνίας του Δουβλίνου. Ενδιαφέρον αυτό, διότι βρισκόμαστε βέβαια μέσα στη μέση των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της Συμφωνίας του Δουβλίνου. Θεωρώ λοιπόν ότι πρόκειται για ένα θέμα όπου πράγματι χρειάζεται να γίνει περισσότερη συζήτηση. Αναμένω βεβαίως με μεγάλο ενδιαφέρον τους επικείμενους τριμήρες διαλόγους. Ευχαριστώ ε, Σίλβια, ευχαριστώ και εσάς κύριε Μακοβέη, λέει ο Πρόεδρος. Είναι σαφές ότι μένει ακόμη δουλειά να γίνει. Είπατε και εσείς άλλωστε ότι υπέρχουν, απέχουν ακόμα τρεις, ε, δύο ε, συναντήσεις τριμερούς διαλόγου και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Ευχαριστώ που μας τα εξηγήσατε αυτά στον διαθέσιμο χρόνο. Θα διακόψω εδώ τώρα την συζήτηση αυτή, διότι σε τρία με τέσσερα λεπτά προβλέπεται η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ και πάλι και όπως είπα ε, υπάρχουν ακόμη δυσκολίες, ευχαριστώ την κυρία Μακοβέη, που μας θύμισε ότι υπάρχουν ακόμα δύο τριμερείς ε, διάλογοι για το θέμα αυτό μέσα στην Εστονική Προεδρία. Ας ε, έχουμε υπόψη ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για ψηφοφορία σε 4 λεπτά και παρακαλώ ελέγξτε αν έχετε τις κάρτες σας.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 Colleagues, uh, we're ready for the vote. Um, just... Συναδελφοί, είστε έτοιμοι. Δεν υπάρχουν συμβιβαστικέ τροπολογίε, οπότε η ψηφοφορία δεν είναι και τόσο εύκολη. Γι' αυτό να προσέχετε τι ψηφίζουμε. Δεν θα πηγαίνω τόσο γρήγορα όσο πηγαίνω συνήθω για να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, είσαστε όλοι προσεκτικοί. Εδώ. Ωραία. Αρχίζουμε. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Θα σας πω περί τίνος πρόκειται για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για μετά το 2020. Η κυρία Μακοβέη είναι η συγκεντριά μας. Κυρία Μακοβέη, θέλετε να πείτε κάτι πριν αρχίσουμε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία μόνο, για τη συνεργασία τέλος πάντων που δεν ήταν πάντα απλή, αλλά νομίζω ότι όλους βοήθησε. Και ελπίζω ότι θα βρούμε τρόπο να καταλήξουμε σε έναν ισορροπημένο Προπολογισμό με ισορροπημένη γνωμοδότηση για τον προπολογισμό, αν μη τι άλλο, για μετά το 2020. Ωραία. Αρχίζουμε με προφορική τροπολογία. Κάπως έτσι, χωρίς να το περιμένουμε, πρέπει να ξέρουμε το περιεχόμενο για να μην ε, βρεθούμε εξαπίνης. Λοιπόν, από το ΕΛΚ είναι η κυρία Μετσόλα, παρακαλώ, να μας παρουσιάσει την προφορική αυτή τροπολογία στην παράγραφο 17. Ευχαριστώ, Κλώτ. Ναι, για να ξέρουμε, όταν μιλάμε για το άρθρο 7, 7 συγγνώμη, 17, 7, τι εννοούμε, ποια είναι η γλώσσα των συνθηκών. Έχει ως εξή. Ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να να επικαλεστεί τη συνθήκη και το κράτος δικαίου στις διάφορες χώρες και ζητάει από το Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του από αυτού. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Λοιπόν, τα ακούσατε όλοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Όχι. Ευχαριστώ. Έγινε. Και διαδικαστικό. Παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν έχω την κάρτα μου, την ηλεκτρονική, οπότε θα ψηφίζω διανατάσσω τη χειρός. Συγγνώμη. Ωραία μας λέτε συν πλήν τέλο πάντων με το χέρι σας για να καταλαβαίνουμε και το προσωπικό εδώ θα καταγράφει την ψήφο σας. Ωραία, όλοι οι υπόλοιποι είσαστε εντάξει με τις κάρτες σας. Πολύ βασικό. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε λοιπόν και αρχίζουμε με την τροπολογία αριθμός 1. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Και άλλος έχει πρόβλημα με κάρτα. Μπορείτε να ψηφίσετε ακόμα. Ψηφίστε. Εντάξει. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 1, δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 4, δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 4, δεύτερο τμήμα. Να παρακολουθείτε, δεν είναι τόσο περίπλοκη η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Τέλειωσε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε. Έτσι καλώ η διαφορά ήταν μεγάλη. Μην ανησυχείτε αν δεν προλάβατε. Ωραία, πιο αργά. Μην τα βάζετε μαζί μου. Τι συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα. Όλοι εντάξει εκεί με το ΕΛΚ, ναι. Ωραία, τροπολογία 2. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 3. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 4. Πρώτο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 τώρα, πρώτο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα της 8. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 9. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 10. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 11. Πρώτο τμήμα. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 11. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 12. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 11, τρίτο τμήμα. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 14 πρώτο τμήμα. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 13. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 15. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 16. Πρώτο τμήμα. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 17. Ψηφίστε παρακαλώ. αλλά εκτός από την τελευταία πρόταση, έτσι, τροπολογία 17 χωρίς την τελευταία πρόταση. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε τροπολογία 17, την τελευταία πρόταση. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. 18. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 19. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 20. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 21. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 23. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 24. Πρώτο τμήμα. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα της 24. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 25. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 26. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. 27. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 28. Ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 29. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 30. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 31. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 32. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 33. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 34. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 35. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 36. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 37. Ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 38. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 39. Ψηφίστε. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. 39. Όχι. Μετά την 38 πάμε στην 41. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 41. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 43 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογίες 44 και 45. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Α, συγγνώμη, απορρίφθηκαν. Όχι, τώρα 46. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος προφορίας. Απορρίφθηκε. 47. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 48. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 51. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της προφορίας. Απορρίφθηκε. 52. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της προφορίας. Απορρίφθηκε. 53. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε 40 ψήφοι υπέρ, 7 κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Τέλειωσε η ψηφοφορία. Και τέλειωσε και η συνεδρίαση. Αν δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα, ωραία καλό βράδυ.